Colleagues, please Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αυτή είναι η τελευταία μας συνεδρίαση για αυτή τη θητεία. Θα προσπαθήσουμε να είναι επιτυχημένη η συνεδρίαση με τόσα πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Να σα θυμίσω ότι όπως συνήθω η συνεδρίασή μας μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο από άψη διερμηνέας έχουμε δώσει προτεραιότητα στις γλώσσε των τακτικών μελών της Υποεπιτροπής Άμυνα και Ασφάλειας. Ας εγκρίνουμε πρώτα την ημερήσια διάταξη. για τη συνεδρίαση αυτή. Αν δεν υπάρχουν σχόλια θα θεωρήσουμε ότι έχει εγκριθεί η μερική διάταξη και σας ευχαριστώ. Θα βρείτε στους φακέλους σας τα πρακτικά των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων. Μία ήταν μια διήμερη συνεδρία 23 και 24 Ιανουαρίου και δεύτερη συνεδρίαση 19 Φεβρουαρίου. έχετε το χρόνο μέχρι το τέλος της σημερινής ε, συνεδρίασης για να υποβάλλετε τυχόν παρατηρήσεις, επιφυλάξεις, ενστάσεις. Οπότε, παρακαλώ, ούτως και πράξτε. Εάν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, θα θεωρήσουμε ότι τα πρακτικά έχουν εγκριθεί. Όσον αφορά τις ανακοινώσεις της Προέδρου, ήθελα να σας πω ότι μετά από το τέλος συνεδρίασης θα θέλαμε να, πάρουμε, να τραβήξουμε μια οικογενειακή φωτογραφία. Δεν βλέπω να είναι πολλά μέλη εδώ παρόντα, αλλά ελπίζουμε να έλθουν περισσότεροι αργότερα. Θα προσπαθήσουμε επίσης να κλείσουμε τη συνεδρίαση με μια εκδήλωση ε, και σας καλούμε να συμμετέχετε όλοι φυσικά. Ας πάμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ε, αφορά τη δημόσια ακρόαση με θέμα τη μεικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την κοινό, ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο. Με μεγάλη μου τιμή Υποδέχομαι τους ε, τρεις διακεκριμένους ε, πανελίστες. Ο πρώτος είναι ο κ. Κόλια Ράουμπε, ανώτατος ε, ερευνητής στο κέντρο πολιτικής κυβερνητικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Λουβένης του Βελγίου στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβένης. Ακολουθεί στη μέση αριστερά μου ο κύριος ε, ο δόκτωρ Hans Born αναπληρωτής ε, συγγνώμη, βοηθός, ε, ε συγγνώμη, υποδιευθυντής στο κέντρο της Γενέβης, ε, στο κέντρο δημοκρατικού ελέγχου των ενόπλων δυνάμεων της Γενέβης. Στη Γενέβη λοιπόν και τέλος ε, ο καθηγητής Κρίστοφερ Λόρντο καθηγητής στο κέντρο Αρένα του Όσλο στην Νορβηγία. Στη διάρκεια της παρουσίας θητείας έχουμε συζητήσει εκτενώς τα γεγονότα που έπονται τα θέματα που έπονται όσον αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα, την ε, κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, ε, την ολοκλήρωση στον τομέα αυτών, το ρόλο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, συζητάμε τη συνολική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και ως επόπτη της διαδικασίας και σε κοινοτικό επίπεδο. με την ταχεία διαδικασία, ειδικότερα κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών. Εξετάζουμε τον ρόλο μας και τη δέσμευσή μας και μαζί με κάποιες σημαντικές εκθέσεις και στις δύο συνεδριάσεις της υποεπιτραπής μας, από κοινού και με άλλες επιτροπές, ειδικότερα την ΑΦΕΤ αλλά και συζητήσεις σε ολομέλειες, σε συνόδους ολομέλειας στο Στρασβούργο και σε μήνυ ολομέλειες στις Βρυξέλλες. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο στους διακεκριμένους πανελίστες. Πρώτος ο, ο Δ. Κόλια Ράουμπ. Ράουμπ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΣΕΝΤΕ, ε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτή την ημερίδα που σημαίνει και την τελευταία συνεδρίαση της, Επιτροπής, της Υποεπιτροπής ΣΕΝΤΕ σε αυτή την ε, θητεία. Η ημερίδα αυτή εστιάζεται σε ένα επίκαιρο ζήτημα, το ρόλο των κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων σε θέματα δημοκρατική λογοδοσία και κοινοβουλευτικού ελέγχου στο πλαίσιο τη ε, πολιτικής, της εξωτερικής πολιτικής και τη πολιτική ασφαλεία. Ένα ε, κλάδο ε, σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι κυβερνήσει. Για να σα δώσω μια γενική επισκόπηση, επέλεξα να δομήσω την παρουσίασή μου ω εξή. Πρώτον, θα εστιαστούμε στο να διευκρινίσουμε στον ορισμό της δημοκρατικής λογοδοσίας, πώς σχετίζεται με την ε, νομιμοποίηση ε, του κοινοβουλευτικού ελέγχου στην ε, εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας πώς τα κοινοβούλια μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες τους για μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία και επιρροή εν ώψη της νομιμοποίησης ουσιαστικά των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. try to. Yes, please. Okay, perhaps I continue. I can, I can change this. Να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια σε λίγο ενώ μεγάλο κομμάτι της συζήτηση επι, επικεντρώνεται στο κοινοβουλευτικό έλεγχο και στην εξέταση. Ε, αναμένεται να δούμε την κοινοβουλευτική νομιμότητα στο πλαίσιο της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. Ας δούμε τη σχέση μεταξύ νομιμότητας και λογοδοσίας της εξωτερικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι, ε, Πολλέ συζητήσει σε ακαδηματικό επίπεδο εστιάζονται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, στην ε, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία. Παρ' όλα αυτά, συχνά είναι ασαφέ πώ αυτά συνδέονται με την δημοκρατική νομιμοποίηση και πώ η δημοκρατική νομιμοποίηση πρέπει να εφαρμόζεται. Σύμφωνα με έναν συναδέλφό μα από το Πανεπιστήμιο του Όσλο, την Ελένη η δημοκρατική εξωτερική πολιτική θα πρέπει να επιδεικνύει ελάχιστη, ένα ελάχιστο δημοκρατική νομιμοποίηση και αυτή η ελάχιστη απέτηση σχετίζεται με τι αρχέ τη αυτονομία και τη λογοδοσία. Δηλαδή η ικανότητα όσων επηρεάζονται από του νόμου να συντάσσουν και τους νόμους αυτονομία και όσοι αποφασίζουν να μπορούν να λογοδοτήσουν για τι αποφάσει του. Και αυτή είναι η λογοδοσία. Όπως γνωρίζουμε σε σχέση με την αρχή της αυτονομίας, η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση θα ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα και η ε, ε, εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφαλείας ε, είναι πολύ λογικό να μπορεί να πει κανεί ότι οι λαοί των κρατών μελών θα πρέπει να εκπροσωπούνται έμεσα από τις κυβερνήσεις τους και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νομιμοποίηση όμως αυτή αφορά πάρα πολλούς παράγοντες θα έλεγε κανείς για να πούμε ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ε, και νομιμοποίηση στις πολιτικές αυτές. Οπότε η αρχή της νομιμοποίησης θα απαιτήσει εναλλακτικέ μορφές εκπροσώπησης ώστε να διασφαλίζεται ότι εκπροσωπούνται εκείνοι οι οποίοι θα επηρεαστούν τελικά από αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα η δημοκρατική νομιμοποίηση απαιτεί ε, τη διατήρηση της αρχής της λογοδοσίας. Δηλαδή, οι αποφάσεις θα πρέπει να ελέγχονται από το νομοθετικό σώμα. Αυτό βασίζεται στην ιδέα ενός κράτους δικαίου, το οποίο επιτρέπει ελέγχους επαναλαμβανόμενους μεταξύ εκτελεστικού και νομοθετικού και απαιτεί μηχανισμούς αυτό εξισορρόπησης της αυτόνομης λήψης αποφάσεων του εκτελεστικού. Με αυτά στο νου μα, αντιλαμβανόμαστε ότι ο ρόλο των κοινοβουλίων στην πολιτική ασφαλεία σχετίζεται κυρίω με αυτό που ονομάζει Vivian Smith ε, νομιμοποίηση ε, στην αρχή, στο τέλος και στη διεξαγωγή. Δηλαδή να υπάρχει διακυβέρνηση από τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους. Ας δούμε εδώ τώρα το ρόλο των κοινοβουλίων στην νομιμότητα και τη λογοδοσία γενικότερα. Μαζί με έναν συναδέλφο από το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου χρησιμοποίησε αυτές τις τρεις ιδέες ε, της ε, ε, input, throughput και output που τα βλέπετε εδώ στο σχήμα. Όταν μιλάμε για το ρόλο των κοινοβουλίων, βλέπουμε το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το πώς συμβάλλουν αυτά σε ε, στη... στοιχεία εισόδου, εξόδου και ε, στην επεξεργασία, στην διεκπαιρέωση της ε, νομιμοποίησης. Και εδώ βλέπετε τι ρόλο παίζουν τα κοινοβούλια και πώ αντιδρούν τα κοινοβούλια με διάφορου τρόπου με την ε, κοινοβουλευτική διπλωματία. Βλέπουμε ότι τα κοινοβούλια συμβάλλουν ενεργά στην ε, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να εστιάζονται στη λογοδοσία και στην έλεγχο. Πώ μπορούν λοιπόν τα κοινοβούλια να επηρεάσουν την ε, εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλεια, επηρεάζοντα τη δημοκρατική αυτονομία και τη λογοδοσία ασκώντα, το να ασκεί κανεί ε, επιρροή δεν περιορίζεται στην ψηφοφορία. Το να ψηφίσει κανεί ε, ή να καταψηφίσει μια πρόταση. Αντί να εστιάζονται αποκλειστικά στη λήψη αποφάσεων, στη φάση δηλαδή της ε, πολιτικής όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις και συμφωνούνται οι αποφάσεις, θα πρέπει να εξετάζουμε και διάφορες άλλες φάσεις της ε, πολιτική λήψη αποφάσεων μαζί με έναν άλλο συναδελφό μου αποφασίσαμε ότι εκεί είναι ουσιαστικά που τα κοινοβούλια μπορούν να κάνουν περισσότερα από ό,τι κάνουν σήμερα. Δηλαδή θα πρέπει να επηρεάζουν και θα μπορούσαν ενδεχομένω να επηρεάζουν το, ε, στάδια λήψη αποφάσεων ε, σε διάφορε περιστάσει. Δηλαδή με άλλα λόγια, θεωρητικά τουλάχιστον τα κοινοβούλια μπορούν να συμβάλλουν στη δημοκρατική λογοδοσία μέσω αυτής της νομιμοποίησης στη φάση, στην ανακτήρια φάση και στην τελική φάση. Ωστόσο, όταν ε, τα κοινοβούλια επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία, είτε την εφαρμόζουν την δημοκρατική λογοδοσία μέσω ελέγχου ή με άλλου τρόπου, αυτό θα εξαρτηθεί από διάφορου παράγοντε. Και πρώτα απ' όλα, οι συναδέλφοί μα από τη Γενέβη, και χαίρομαι που ο Χανσπόρ είναι εδώ, μα έχουν δείξει σε πολλέ μελέτε ότι αυτό εξαρτάται από τι ε, επίσημε εξουσίε, την εξουσία των κοινοβουλίων, τι δυνατότητε, τι ικανότητέ του, αλλά και κυρίως από την βούλησή τους. Δεύτερον, διάφοροι παράγοντες ε, ε, του περιβάλλοντος ε, επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας των κοινοβουλίων. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη νέων κοινοβουλευτικών συνθήκων που επισημοποιούν ορισμένες πρακτικές και ορισμένους κανόνες. Ας δούμε το Ηνωμένο Βασίλειο για αυτό η παράκαμψη των κοινοβουλίων μέσω ε, εκτελεστικής δράσης, δράσεων του εκτελεστικού είναι ένα άλλο μέσο και τέλος η πολιτικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας παραμένει σημαντικός παράγον που εξηγεί γιατί τα κοινοβούλια θα έπρεπε να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και βούληση να χρησιμοποιούν όχι μόνο την εξουσία και την ικανότητά τους, αλλά ε, και να προωθούν ε, τη βούλησή τους στον τομέα. Ποια είναι η επίδοση τη δημοκρατική λογοδοσία και του ελέγχου, τι μορφή θα έχει αν εξετάσουμε τι βασικέ ε, κοινοβουλευτικέ λειτουργίε ω ε, μηχανισμό ελέγχου, εξέταση, ε, λήψη αποφάσεων, νομοθεσία και κοινοβουλευτική διπλωματία. Πρώτα απ' όλα μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ κοινοβουλευτικού ελέγχου αφενό και κοινοβουλευτική εξέταση από την άλλη. Ο κοινοβουλευτικό έλεγχο συνεπάγεται εξουσία κύρωσης του εκτελεστικού βέτο, δηλαδή ε, ακύρωσης αποφάσεων. Οι εξουσίες κοινοβουλευτικού ελέγχου δίνει τη δυνατότητα θέσης βέτο στο εκτελεστικό σε ε, περίπτωση ας πούμε δημοσιονομικών θεμάτων ε, ή νομοθετικών θεμάτων ή θεμάτων που αφορούν πόλεμο. Η εξέταση αφορά πιο ήπια κοινοβουλευτικά μέτρα για να καλούνται προλογοδοσίες ορισμένοι εξωματούχοι Η εξέταση ε, απαιτεί διαβούλευση του Κοινοβουλίου στη χάραξη πολιτική και τα κοινοβούλια μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εξουσία του κόσμου, του λαού, για να εξετάσουν νομοθετικέ πράξει, ε, να νομιμοποιήσουν ή να τι απονομιμοποιήσουν ενώπιον του λαού. Μάλιστα, σε ορισμένε περιπτώσει, κάποιε κυβερνήσει ζητούν εξέταση κοινοβουλευτική ώστε να νομιμοποιήσουν τι δράσει του δημοσίω. Τρίτον, τα κοινοβούλια μπορούν ε, να λαμβάνουν αποφάσεις και να νομοθετούν, για παράδειγμα, σε σχετικούς τομείς πολιτικής και συνεπώς έμεσα να επηρεάζουν ε, τον έλεγχο και την εξέταση της ε, κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας και μετά προστίθε άλλο ένα επίπεδο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Ας δούμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήδη το 1990 ο Ρόλαντ Μπίπερ ισχυρίστηκε ότι η εμπλοκή του Κοινοβουλίου είναι αναγκαία για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του συστήματο χάραξη εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερο χρειάζεται να λαμβάνει πολύπλοκε αποφάσει. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλε οι, οι οπτικέ γωνίε πολιτική ε, και του Κοινοβουλίου. Αυτό συζητήθηκε το 1990 ήδη. Σήμερα, ακόμα σήμερα ορισμένοι συντάκτες στηρίζουν, υποστηρίζουν ότι η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ε, ασφάλειας και η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ε, ε, πρέπει να έχουν και τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, η κύρια εξουσία ανήκει σε άλλους στους εκτελεστικούς φορείς όπως το Συμβούλιο, στην ύπατη εκπρόσωπο και στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Επίση, θα μπορούσε κανείς να πει ότι μετά από τη Λισαβόνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, κέρδισε περισσότερες εξουσίες όχι μόνο όσον αφορά τη λογοδοσία του στην ε, κοινή πολιτική ε, ασφαλείας και άμυνας αλλά και ω σημαντικός φορέας σε διεθνεί σχέσει. παρά το σχετικά περιορισμένο επίσημο ρόλο στην CSDP έχουν βρεθεί άτυπε διευθετήσει που βαθμία ενισχύουν τον σχετικά περιορισμένο ρόλο όπως γνωρίζετε συμπεριλαμβάνουν και την δήλωση πολιτικής λογοδοσίας, ε, πρόσβαση σε έγγραφα και σε ακροάσεις ε, αντιπροσωπιών, απλά για να πούμε ορισμένα. Ε, ταυτόχρονα, πιο ουσιαστικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επηρέασε τη χάραξη και τη δόμηση της, εξωτερικής, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, την παγκόσμια στρατηγική και πιο πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο για να επηρεάσουμε. Επιστρέψουμε στο θέμα της ε, επιρροής του ΚΕΠΑ. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι άτυπες εξουσίες ε, σχετίζονται με την επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διάφορες φάσεις χαραξής πολιτικής, τόσο όσον αφορά πριν τη λήψη αποφάσεων, όσον αφορά και τη διαδικασία λήψη αποφάσεων, αλλά και μετά από τη λήψη αποφάσεων. Κοιτώντα τώρα την υπόθεση των Εθνικών Κοινοβουλίων στην πολιτική ασφαλεία, βλέπουμε πολλέ διαφορετικέ παραλλαγέ όσον αφορά ε, τι εξουσίε, την νομοθετική, δημοσιονομική και ε, εποπτική εξουσία ε, σε διάφορε χώρε. Αυτό σχετίζεται κυρίω με τι εξουσίε που αφορούν θέματα πολέμου, ε, και βλέπουμε μια διαφορά ε, μεταξύ κοινοβουλίων που έχουν εξουσίε ε, βέτο εκ των προτέρων και που δεν, των άλλων που δεν έχουν, αλλά έχουμε και άλλα κοινοβούλια που έχουν πρόσφατε εξουσίε ε, ή που έχουν χάσει πρόσφατα εξουσίες. Ε, κάποια κράτη-μέλη έχουν αλλάξει τι εξουσίε αυτέ μετά από τον πόλεμο στο Ιράκ. Αλλά αναβάθμισαν το ρόλο των κοινοβουλίων και άλλα τον υποβάθμισαν ε, δεδομένου ότι πρόκειται να, να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Το 2018 το, η Βουλή των Κοινοτήτων καταψήφισε την εμπλοκή Βρετανικών δυνάμεων στη Συρία. Αυτό οδήγησε κάποιους συναδέλφους να λένε ότι ουσιαστικά βλέπουμε ε, μια νέα άτυπη σύμβαση ε, να εμφανίζεται στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Αυτές οι συγκριτικές ε, διαπιστώσεις οδηγούν συναδέλφους στο να αναφέρονται ότι υπάρχει μια τάση περισσότερης εμπλοκής των κοινοβουλίων ή λιγότερης ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα ισχυρίζεται ότι η θεωρία της δημοκρατικής ειρήνης ε, μπορεί ακόμα να ισχύει όσον αφορά την, το κατά πόσο πάμε σε πόλεμο, πάει μια χώρα σε πόλεμο ή όχι. Δεδομένων αυτών μπορούμε να πούμε συνολικά ότι το πόσο επηρεάζει ένα κοινοβούλιο τα πράγματα εξαρτάται από το πόσο ένα κοινοβούλιο επηρεάζει την κατάσταση ασφαλείας. Δύο ε, ζητήματα τίθενται. Σε εθνικό επίπεδο βλέπουμε εκτεταμένη συνένεση των κοινοβουλίων για θέματα πολέμου παρά τα συστήματα με λιγότερε εξουσίε για το κοινοβούλιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ερώτημα είναι, θα δούμε να υπάρχει μεγαλύτερη κοινοβουλευτική επιρροή ε, στο πλαίσιο μη τυπικών εξουσιών. Τέλος, θα πρέπει να εξετάσουμε το ρόλο της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας ως γέφυρας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτέ οι πολιτικέ ασφαλεία και άμυνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΚΕΠΑ, μπορούν να αποτελέσουν μια στρώση ανταλλαγή πληροφοριών και όχι μόνο, αλλά και για την ανταλλαγή μηχανισμών λογοδοσία στο πλαίσιο τη ΚΕΠΑ. Και τέλο, πώ ο διευρυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την κοινοβουλευτική διπλωματία θα μπορούσε να βοηθήσει όχι μόνο για να ενδυναμωθούν οι ευρωπαϊκές δράσεις επιτόπου, αλλά και για την ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας. Πριν κλείσω, θα ήθελα να σας πω τα εξή. Προσπάθησα να απαντήσω το ερώτημα που αφορά το ρόλο των κοινοβουλίων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Δηλαδή, τι ρόλο παίζουν σε θέματα δημοκρατική λογοδοσία και κοινοβουλευτικού ελέγχου σε ζητήματα πολιτική ασφάλεια. Με την ανάγκη μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία εν ώψη ε, ε, σταδίων και των τελικών σταδίων της δημοκρατικής λογοδοσίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η σύγκρισή τους μας οδηγούν στο ερώτημα του ποιο στο μέλλον θα νιώσει την νομιμοποίηση της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής σε αυτό το τομέα. Χρειάζεται περισσότερη συμμετοχή των κοινοβουλίων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαφορετικά θα ζήσουμε κοινοβουλευτικό έλλειμμα στην ΚΕΠΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Dr. Ε, Hans ε, Born, ε, υποδιευθυντή της DCAF στην Γενέβη. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση να είμαστε ανάμεσά σας. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, είναι λίγο πολύ. Ε, η τελευταία μέρα για αυτή την Επιτροπή, στη συνέχεια όλοι μας τον Μάιο θα πάμε να ψηφίσουμε και θα ε, συσταθεί νέο κοινοβούλιο στη συνέχεια τον Ιούνιο και 2 Ιουλίου, αρχές ε, Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι νέες επιτροπές. Ε, βλέποντας λοιπόν απ' έξω την ε, κατάσταση και αυτό είναι το οποίο θα ήθελα να συζητήσω και μαζί σας είμαι λίγα και διότι άμα δούμε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες έχουν μια πλήρη επιτροπή σχετικά με τις αμυντικές πολιτικές κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι το οποίο είναι περίεργο. Είναι υποεπιτροπή εδώ. Είναι σημαντικό, δεν θέλω να υποτιμήσω ε, την αξία της. Ε, όμως ε, πιστεύω ότι εν ώψην όλων αυτών τα κράτη-μέλη εργάζονται όλο και πιο στενά στο πλαίσιο της ΠΕΣΚΟ αυτήν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε ζητήματα άμυνας έχουμε 35 συνολικά προγράμματα που πραγματοποιούνται και φυσικά ποιο θα τα επιβλέπει. Μια επιτροπή ναι μπορεί να το κάνει, όμω μια πλήρη επιτροπή θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη δικαιοδοσία για κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο. Το δεύτερο είναι ότι η άμυνα και η ασφάλεια για την Ευρώπη θα παραμείνει μια υψηλή προτεραιότητα, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Βλέπουμε γύρω από την Ευρώπη μια ζώνη αστάθειας ε, στην Ουκρανία, στη Μεσόγειο, ε, στην Ουκρανία έχουμε την ε, Ρωσία που έχει μια ιδιαίτερα επιθετική στάση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει αποστείλει στρατεύματα στο εξωτερικό και τέλος τι γίνεται με την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αμυνθεί τον εαυτό της όταν ουσιαστικά οι Ηνωμένε Πολιτείε περιορίζουν τις εξουσίες τους. Έχουμε αυτή τη στιγμή έναν πρόεδρο ο οποίος ε, έχει μια τέτοια ε, θέση. Οπότε μπορούμε να βασιζόμαστε ακόμα στις Ηνωμένε Πολιτείε όπως κάναμε και τις προηγούμενες δεκαετίες. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δημιουργήσει δηλαδή μια στρατηγική αυτονομία ούτω ώστε να φροντίσει την ίδια της την ασφάλεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουν οι πολίτες της Ένωσης από την Ένωση. Και αυτά ήθελα να δηλώσω ε, ως ένα εισαγωγικό πλαίσιο. Και τώρα θα περάσω στην ε, σύντομη παρουσίασή μου Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά είναι τεχνικά όμως βρισκόμαστε σε ένα πολιτικό κοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν ε, να το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Έτσι λοιπόν για σήμερα θα επικεντρωθώ ε, για στα κοινοβούλια των ε, κρατών μελών σχετικά με την εξωτερική του άμυνα και στη συνέχεια Ε, τι γίνεται όσον αφορά την αποστολή στρατευμάτων στο εσωτερικό των χωρών. Αρχικά λοιπόν θα ήθελα να σας πω ποιοι είμαστε το DCAF, τι οργανώσεις είμαστε. Είμαστε ένας ε, διεθνής οργανισμός με 65 μέλη, όλα τα κράτη-μέλη είναι ε, μέλη μας και προωθούμε την καλή διακυβέρνηση του τομέα ασφάλειας. Προωθούμε δηλαδή αποτελεσματική ε, άμυνα η οποία όμως και λογοδοτεί. Κατά 75% είμαστε λειτουργικός οργανισμός, κάνουμε δραστηριότητες κατά τόπους, με κυβερνήσεις, με χώρους, ώστε να ενισχύσουμε τη διακυβέρνηση του δικού του τομέα άμυνας. Ε, μπορούμε να τους υποστηρίξουμε, δεν αναλαμβάνουμε πλήρως ε, την ε, δράση αυτή και επίσης είμαστε και μια δεξαμενή σκέψη και αυτό είναι το κομμάτι στο οποίο εργάζομαι εγώ και έτσι θα σας παρουσιάσω ένα κομμάτι του έργου μας. Τώρα, άμα δείτε τις βασικές στατιστικές, έχουμε, 100, ε, έχουμε 65 κράτη-μέλη, έχουμε συνολικά 160 άτομα προσωπικά, 40 ε, εθνικότητες ε, και έχουμε δράσει σε 70 χώρες. Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρισκόμαι σήμερα εδώ. Έχουμε εργαστεί με συνεργαστεί και στο παρελθόν με την Επιτροπή ΣΕΝΤΕ και χαιρόμαστε ιδιαίτερως για αυτό. Η Επιτροπή ΣΕΝΤΕ δεν είναι η μόνη. Έχουμε συνεργαστεί και με την ΛΥΜΠΕ, με την ε, Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων, Και τώρα περνάω στην παρουσίαση. Όπως είπα θα επικεντρωθώ σε δύο τομείς, ε, στις στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό, καθώς επίσης και την ε, χρήση ε, στρατιωτικών αποστολών στο εσωτερικό. Και αυτό βασίζεται στο έργο το οποίο έχουμε διεξαγάγει. Αρχικά λοιπόν δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Άμα δούμε όμως τι κάνουν ακριβώς τα κοινοβούλια μπορούμε να ε, χωρίσουμε το έργο τους ε, σε πέντε τομείς. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ε, κάνουν, έχουν κοινοβουλευτικό έργο, κάτι το οποίο κάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ελέγχουν επίσης τον προϋπολογισμό, έχουν την επίβλεψη, κάνουν ελέγχους, έχουν αντιπροσωπευτικό ρόλο, κάνουν συζητήσεις, ενημερώνουν τους πολίτες και φυσικά έχουν και εκλεκτικό ε, ρόλο εκλογής, δηλαδή ορίζουν ε, ε, τους επικεφαλείς σε διάφορες υπηρεσίες. η επί... το... αυτόν τον ρόλο το βλέπουμε και εδώ στο Κοινοβούλιο όπου οι επίτροποι θα πρέπει να περάσουν από εδώ ε, να ε, μιλήσουν ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι επίσης ένας από τους ισχυρότερους ελέγχους που κάνει το Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαίτερως όσον αφορά τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με αυτές τις πέντε εξουσίες δεν είναι ισότιμα διανεμημένες μεταξύ των... στα διάφορα κράτη-μέλη και θα μιλήσω ε, με το παράδειγμα των αποστολών στο εξωτερικό. Το δεύτερο θέμα τώρα είναι ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το τριπλό αλφα των κοινοβουλίων είναι ε, ένα πλαίσιο το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς ε, στη δουλειά μας. Δεν θα πρέπει να εξετάσουμε τις επίσημες εξουσίες ε, των κοινοβουλίων ή τα μεγαλακτήρια όπου βρίσκονται. Από τη μία έχουμε τις νομικές εξουσίες που δίνονται στο κοινοβούλιο. Επιτρέπεται λοιπόν να έχουν λόγο για την αποστολή στρατογμάτων στο εξωτερικό. Δεύτερον έχουμε τους πόρους οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών και τέλος έχουμε την στάση. Τι κάνουν δηλαδή τα διάφορα οι διάφοροι βουλευτές πάνω σε αυτό το θέμα. Βλέπουμε ότι σε όλες τις χώρες, ακόμα και σε αυτές με τις περισσότερες ε, εξουσίες, ε, οι ε, βουλευτές δεν θέλουν να βάλουν την κυβέρνηση τους να λογοδοτήσει γιατί ανήκει στο ίδιο κόμμα με τους ίδιους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να εξετάσουμε τις μεμονωμένες ε, θέσεις των κοινοβουλίων και των βουλευτών. Ε, βέβαια μπορούμε να πούμε ότι εξαρτάται από τον κάθε βουλευτή, διότι και αυτοί έχουν μεγάλη πίεση από, τους, από το κόμμα τους να ψηφίζουν με βάση τη γραμμή του κόμματος. Δεν είναι κάτι μεμονωμένο, θα πρέπει λοιπόν να το δούμε σε έναν πιο διαρθρωμένο τρόπο. Τώρα όσον αφορά τις αποστολές στο εξωτερικό, εάν το δούμε συγκριτικά, ο μεγαλύτερος πάροχος αποστολών είναι τα Ηνωμένα Έθνη με πάνω από 100.000 προσωπικό. Μετά έχουμε το ΝΑΤΟ με 6 αποστολές και 20.000 προσωπικό και τέλος έχουμε ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση με 6 αποστολές και 4.000 άτομα προσωπικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από οικονομική άποψη από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στον πλανήτη, όμως μία από τις μικρότερες όσον αφορά το το στρατιωτικό κομμάτι και έτσι λοιπόν φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζεται πιο γι' αυτόν τον λόγο ε, ως μια ήπια δύναμη. Δεν θα πρέπει να μιλάμε μονάχα για στρατιωτικές αποστολές, διότι πολλές αποστολές ε, σήμερα είναι μικτές ε, με αστυνομικούς, με δικούς που ε, μπορούν να βοηθήσουν στην οικοδόμηση των κοινωνιών. Είναι μια μεικτή κατάσταση λοιπόν. Εάν εξετάσουμε λοιπόν την κατάσταση για αυτόν, οι πέντε βασικές χώρες ε, που, συμμετέχουν σε, που συνεισφέρουν στις αποστολές δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική μου χώρα, οι 100 χώρες, ε, είναι μία από τις ε, πιο σημαντικές χώρες οι, περισσότεροι, οι περισσότερες περιπτώσεις λογοδοσίες γίνονται σε εθνικό επίπεδο και όχι σε διεθνές επίπεδο και θα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό λοιπόν ε, εάν ε, όσον αφορά τις χώρες που συνεισφέρουν όπου είναι η Αιθιοπία, η Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και ούτω καθεξής. Και τώρα θα ήθελα να επικεντρωθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στο κίτρινο θα πρέπει να εξετάσουμε την στιγμή που γίνεται η αποστολή των στρατευμάτων. Από εκεί τα κοινοβούλια μπορούν να παίξουν έναν ρόλο. Θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν τις διάφορες φάσεις της λήψης αποφάσεων. Αρχικά έχουμε την ε, κοινή δράση του Συμβουλίου όπου αποφασίζεται ότι θα στείλουμε. Στη συνέχεια το κράτος μέλος αποφασίζει να συμμετάσχει σε αυτή την αποστολή και στη συνέχεια έχουμε τα στρατεύματα κατά τόπου. Θα εξηγήσω στη συνέχεια ότι πολύ συχνά επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στη στιγμή όπου τα στρατεύματα ε, φτάνουν στην τοποθεσία τους και τότε είναι ήδη πολύ αργά. Βλέπουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να χωρίσουμε τα κοινοβούλια της Ένωσης σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με την συμμετοχή τους. Υπάρχουν κάποιες χώρες όπου υπάρχει προέγκριση πριν από την διεθνή απόφαση, δηλαδή πριν το, την, απόφαση του, ε, του κοινού, την κοινή απόφαση του Συμβουλίου. Στη συνέχεια υπάρχουν ε, χώρες που γίνεται έγκριση αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να αποστείλει στρατεύματα Όμω πριν από την εθνική απόφαση, στη συνέχεια υπάρχουν χώρες που έχουν συμβουλευτικό ρόλο, όχι αποφασιστικό ρόλο όμως, και τέλος υπάρχουν κοινοβούλια τα οποία δεν έχουν πραγματική εξουσία σε αυτόν τον τομέα. Αυτά τα παραδείγματα λοιπόν δεν είναι σχετικά. Αυτό το οποίο θα ήθελα να, να, στο οποίο θα ήθελα να επικεντρωθώ είναι ότι χώρες οι οποίες ε, βρίσκονται, υπάρχουν χώρες όπου έχουν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση όπου έχει ληφθεί μια απόφαση ήδη εδώ στις Βρυξέλλες. Έχουμε χώρες όπου η Γερμανία, οι κάτω χώρες όπου η κυβέρνηση έρχεται εδώ στις Βρυξέλλες, επιστρέφει στην πρωτεύουσα και στη συνέχεια λέει στο κοινοβούλιο «Ωραία, συμφωνήσαμε στις Βρυξέλλες ότι θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό» κτλ. κτλ. Θα πρέπει να δράσουμε τώρα και θα πρέπει να συμφωνήσετε διότι η δάλωση, η φήμη μας ε, διακυβεύεται. Βλέπετε λοιπόν ότι πολύ συχνά τα κοινοβούλια αυτά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο παρά μόνο να ακολουθήσουν την απόφαση της κυβέρνησης. Οπότε θα πρέπει να, για να έχουμε πραγματική επίβλεψη τα κοινοβούλια να λαμβάνουν μια απόφαση πριν λάβει απόφαση το Συμβούλιο. θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι ανάγκη, η κυβέρνηση είναι αυτή που κυβέρνει, οπότε, που κυβερνεί, οπότε αυτή παίρνει την απόφαση. Εάν το Κοινοβούλιο είναι να παίζει μεγαλύτερο ρόλο, θα πρέπει να εξετάσουμε τη στιγμή όπου το Κοινοβούλιο αναλαμβάνει δράση. Έχουμε βρει κάποια πρακτικά παραδείγματα σχετικά με το πώς το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει αυτές τις αποστολέ Κάποιες χώρες όπως η Σουηδία θα πρέπει να δημιουργήσουν, να ψηφίσουν μια ειδική νομοθεσία για κάθε αποστολή. Στη συνέχεια έχουμε τη Φινλανδία εάν ένας ε, υπουργό πάει στις Βρυξέλλε να διαπραγματευτεί μια τέτοια απόφαση του Συμβουλίου, πριν πάει θα πρέπει να εξηγήσει στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ε, το ποια θα είναι η θέση τη Φινλανδίας στην προκειμένη περίπτωση και τρίτον έχουμε ε, πολύ ενδιαφέρον εδώ πέρα τα περισσότερα συντάγματα είναι πολύ παλιά συντάγματα των κρατών μελών και επικεντρώνονται κυρίως ε, στις ένοπλες δυνάμεις και όχι στην αστυνομία. Οπότε ακόμα και αυτές οι χώρες δεν προσέχουν ιδιαιτέρως ε, στο ζήτημα της αποστολής της αστυνομίας στο εξωτερικό. Εξαίρεση τώρα είναι το Λουξεμβούργο, η Σουηδία, η Φινλανδία που λένε δεν κάνουμε διάκριση σχετικά με το αν είναι κάποιος στρατιωτικός ή αστυνομικός. οποιοδήποτε. Ε, μπορεί να χρησιμοποιήσει ε, εξουσία, δύναμη, ε, θα πρέπει να ελέγχεται από το Κοινοβούλιο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι πολύ πολύπλοκο. Θα το αφήσουμε στην κυβέρνηση και εμεί απλά θα ακολουθήσουμε την κυβέρνηση. Είναι μια πολιτική απόφαση που θα πρέπει να, να την λαμβάνουν σε κάθε κράτος μέλος. Αυτό αφορά τον τρόπο αποστολής στρατευμάτων. Τώρα θα ήθελα να πω την χρήση ε, δυνάμεων στο εσωτερικό μιας ε, χώρας. Ο εσωτερικός ρόλος ε, των ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από δύο αρχές. Από τη μία έχουμε την αναλογικότητα. Κάθε δράση θα πρέπει να είναι ανάλογη της ασφάλειας και η επικουρικότητα θα πρέπει να υποστηρίζει τις εθνικές αρχές θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι διαφωνούν με κάτι τέτοιο. Έχουμε λοιπόν τρεις, τρεις τύπους εσωτερικών ρόλων ε, την διατήρηση της δημόσιας τάξης, ε, περίπτωση φυσικής καταστροφής ε, και ρόλος που δεν σχετίζεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια. Για παράδειγμα, σε ορισμένες χώρες η όταν γίνεται απεργία των ε, απορριμματοφόρων για πολλές εβδομάδες, η κυβέρνηση αποφασίζει ότι το ρόλο αυτό θα πρέπει να τον αλάβει ο στρατός. Κάτι το οποίο έχει γίνει κάποτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η χρήση των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό σχετίζεται πάντοτε με έκτακτες συνθήκες και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι εδώ έχουμε την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ κοινοβουλίου και της εκτελεστικής εξουσίας αλλά και με το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό το οποίο βλέπουμε λοιπόν σχετικά με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι τα περισσότερα κοινοβούλια ε, αναμειγνύονται όταν γίνεται μια τέτοια, είναι να ληφθεί μια τέτοια απόφαση. Όμως το ενδιαφέρον είναι ότι οι μισές, τα μισά κράτη-μέλη δεν έχουν ε, μια, ε, έναν κανονισμό σχετικά με την επιμήκυνση, την ολοκλήρωση αυτής της απόφασης. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κράτη-μέλη που είναι πολύ αυστηρά σχετικά με το πώς θα ξεκινήσουν μια κατάσταση εκτέκτου ανάγκης, όμως δεν ισχύει το, το ίδιο σχετικά με τη λήξη αυτής. Και ολοκληρώνοντας την παρουσίασή μου τώρα, είπα ήδη στην αρχή ότι η άμυνα και η ασφάλεια είναι μια υψηλή προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να δούμε αυτά τα θέματα σε διάφορα επίπεδα, όπως, όπως για παράδειγμα η αύξηση της συνεργασίας, ειδικά ζητήματα όπως η καταπολέμηση του εξτρεμισμού, η μετανάστευση ή και θέματα όπως είναι για παράδειγμα η επίβλεψη των ειδικών δυνάμεων, ε, των μυστικών υπηρεσιών και θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ κύριε και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον καθηγητή κύριο Κρίστοφερ Λόρντ, καθηγητή του Κέντρου Αρένα στο Όσλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Θα σας πω ευθύς εξ αρχής ότι ελάχιστα γνωρίζω για θέματα άμυνας και ασφάλειας. Δραστηριοποιούμε κυρίως ε, για αφηρημένα φιλοσοφικά ζητήματα δημοκρατικότητας και ε, νομιμοποίησης, ε, αιτιολόγησης δηλαδή της πολιτικής δύναμης. Οπότε προσπαθώ να καταλάβω ε, και να, εφαρμό, να δω πώς καταλαβαίνουμε και εφαρμόζουμε αυτές τις βασικές αρχές της πολιτικής και στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με αυτό το υπόβαθρο θα σας πρότεινα πέντε αιτίες για τις οποίες πιστεύω εγώ ότι η κοινοβουλευτική συμμετοχή στην πολιτική ασφαλείας είναι ουσιώδου σημασίας και γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχει σε αυτό το μείγμα με τα εθνικά κοινοβούλια, όπως εννοείται. Πρώτον, η ευρωπαϊκή πολιτική ασφαλείας ε, απαιτεί συντονισμό των εξουσιών και των ικανοτήτων των κρατών μελών Προφανώς αυτή η πολιτική ε, ωστόσο γίνεται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμφωνίες ε, επιτυγχάνονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο των Υπουργών. Τα κράτη-μέλη συχνά αποφασίζουν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες και τις γνώσεις της Κομισιόν όσον αφορά την, ε, το σχεδιασμό της εξωτερική εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας ή της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας οι δηλώσει ε, σε θέματα ασφάλεια, οι δράσει, οι αποστολέ γίνονται εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικαλούνται την εξουσία τη ε, και ρηψοκινδυνεύουν την αξιοπιστία τη. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει δυνάμει εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αν αυτέ οι δυνάμει είναι δυνάμει των κρατών μελών. Και σε αυτή την περίπτωση η δράση αυτή ρίψο κινδυνεύει την αξιοπιστία και τη φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποστολές αυτές επικαλούνται ευρωπαϊκές αξίες, αιτιολογούνται συχνά ε, με την πρόθεση των ευρωπαϊκών αξιών. Οι αποστολές ασφαλείας αποστέλλονται ε, βάσει εντολών που έχουν συμφωνηθεί από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, φέρουν τις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν τη φήμη και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασφάλειας και συνεργασίας, τότε αυτή η συνεργασία σε θέματα ασφάλειας θα πρέπει να λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, η δημιουργία ε, δυνάμεων ασφαλείας μέσα στο χρόνο απαιτεί στοιχήματα, κινδύνους απαιτεί κοινοβουλευτική συμμετοχή μέσα στο χρόνο η οποία παρέχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσω ενός συνδυασμού εθνικής συμμετοχής και ευρωπαϊκής συμμετοχής, εθνικών και ευρωπαϊκών ε, κοινοβουλίων και ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Σκεφτείτε μια ολόκληρη σειρά ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών σε θέματα ασφάλειας, πράγματα που έχουν γίνει πραγματικά, που συνέβησαν ήδη πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή για να βρείτε ιδέες για το μέλλον. Φανταστείτε μια ευρωπαϊκή δύναμη ταχείας ε, ε, επέμβασης, ε, μάχημες δυνάμεις, έναν οργανισμό εξοπλισμών που θα προωθεί τις ικανότητες και τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων, τη συγκέντρωση και ομαδοποίηση συγκεκριμένων δυνάμεων, όπως συγκέντρωση πληροφοριών. Και φυσικά συνεργασία διαρθρωτική. Ανέφερε ο Χάνς τις πέντε πρωτοβουλίες και που θα μας οδηγούσαν σε μια καλή διαρθρωτική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών που θέλουν να ενοποιήσουν τις δυνάμεις τους περισσότερο από τι άλλες. Όσο μεγαλύτερη είναι η ομαδοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας, τόσο περισσότερο απαιτείται κατανομή των καθηκόντων και τόσο πιο δύσκολο θα είναι για επιμέρους κρατημέλη να επιστρέψουν στην αυτάρκεια σε θέματα ασφάλειας. Όσο μεγαλύτερη είναι η συνεργασία, όσο μεγαλύτερος είναι ο συντονισμός στην ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων τους, τόσο πιο δύσκολο είναι να πάνε πίσω ή να επιχειρήσουν στο να πάνε πίσω στην αυτάρκεια, ε, να παρέχουν δηλαδή τις δικές τους δυνάμεις μόνοι τους, μόνα τους. Ε, οπότε κάθε απόφαση κατανομής ε, των καθηκόντων, εξειδίκευση, συντονισμού μέσα στον χρόνο είναι ένα στίχημα, ένας κίνδυνος. Είναι ένα στίχημα που μπορεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία των άλλων, των εταίρων, την αξιοπιστία των άλλων κρατών μελών. Θα τα καταφέρουν, θα βρίσκονται εκεί, θα μας συνδράμουν όταν θα χρειαστεί, θα συμμετέχουν πράγματι σε ε, αποστολές όταν αυτό χρειαστεί. αλλά και οι αποφάσει μη συνεργασία είναι στοιχήματα. Με όποιον τρόπο και να το σκεφτεί κανεί, τα κράτη-μέλη στοιχηματίζουν την αξιοπιστία του όταν αποφασίζουν να συνεργαστούν σε θέματα άμυνα, αλλά και όταν αποφασίζουν να μη συνεργαστούν. Είναι το στοίχημα τεράστιο. Σε έναν κόσμο γεμάτο κινδύνου, όπου τα, κάθε κράτο μέλο ελάχιστα μπορεί να κάνει για την ασφάλεια, το ακόμη και ένα μεγάλο κράτο μέλο, ο κίνδυνο τη μη συνεργασία μπορεί να είναι το ίδιο μεγάλος όσο και αυτός της συνεργασίας. Όποια και αν είναι η επιλογή θα υπάρχουν κίνδυνοι. Οπότε όσο όλο και περισσότερο οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποιούνται βάσει το δεδομένου ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιηθούν μαζί με εταίρου, τόσο περισσότερο θα πρέπει να εμπλακούν αξιόπιστα και εκ των προτέρων τα κράτη-μέλη. Εξού και αυτό το σημείο κλειδί που ανέφερε ο Χάντς δεν έχει νόημα να εκφράζονται δεσμεύσεις ε, για δυνάμεις ε, πριν τις κρίσεις τα, τα, ε, θα πρέπει να γίνονται όλες αυτές οι δεσμεύσεις και οι συνεργασίες εκ των προτέρων θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία δεσμεύση μεταξύ εταίρων για να μπορούν να συνεργαστούν, θα μπορούν να επωφεληθούν από κάποιο είδους ε, ε, διαρκείς διαβουλεύσεις, ε, διαρκή διάλογο για τα πρότυπα, τις αξίες και τα δικαιώματα που αιτιολογούν αυτή την ομοδοποίηση ε, δυνάμεων. Και αυτόν ακριβό το ρόλο παίζουν τα κοινοβούλια. Θέτουν τα πρότυπα, τα δικαιώματα και τις αξίες. Τέτοιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε ένα δημοκρατικό σύστημα από κοινοβούλια επιχειρησιακές και τεχνικές αποφάσεις ε, μπορούν να λαμβάνουν και οι κυβερνήσει. αλλά το πρότυπα, τα δικαιώματα και οι αξίες πρέπει να αποφασίζονται βάσει ευρωπαϊκής συνεργασία από τα κοινοβούλια. Και όπως είπα, πρέπει να αποφασίζονται μέσω ενός διαρκούς διαλόγου που θα γίνεται πριν ξεσπάσουν οι κρίσει, ώστε τα κρατημένα να μπορούν να συνεργαστούν αξιόπιστα μεταξύ του, για να ε, αναπτύξουν όλες αυτές τις δυνατότητες. Πρώτον, η συνεργασία σε θέματα ασφάλειας είναι ένα διεθνές ε, κοινοφιλές αγαθό. Με άλλα λόγια, τα κράτη-μέλη από μόνα τους ε, είναι δύσκολο να ξερουμε συγκεκριμενα συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Αν αυτό συμβεί, αν είναι να έχουμε συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, είναι δύσκολο να εξαιρεθούν από αυτά τα ωφέλη κάποια κράτη-μέλη. Οπότε πώς μπορεί να διασφαλίσει κανείς ότι κάποια κράτη-μέλη δεν θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τη συνεργασία, εποφελούμενα από αυτήν, χωρίς να συμβάλλουν με το απαραίτητο κόστος. Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι κάποια κράτη-μέλη δεν θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν αρνητικούς εξωτερικούς παράγοντες ε, το ένα στο άλλο. Σκεφτείτε ένα κράτος μέλος, για παράδειγμα, το οποίο ε, βγάζει τεράστια χρήματα από έναν τεράστιο χρηματοπιστωτικό τομέα, ε, στον οποίο παρατηρείται ξέπλυμα χρήματος εκτενές, αυτό επηρεάζει ως εξωτερικός παραγόν άλλα κράτη-μέλη. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν. Ε, η δυσκολία είναι να δούμε κατά πόσο αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, κάποια κράτη-μέλη να ε, ε, εκμεταλλευτούν την ασφάλεια που παρέχεται με αυτόν τον τρόπο εις βάρος ή κάποια, αν κάποια κράτη-μέλη θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν κάποιους εξωτερικούς παράγοντες σε άλλα. Εάν τα εν λόγω κράτη-μέλη έχουν συμφέρον να κάνουν αυτά τα κακά πράγματα, τότε μιλάμε για εκδείξη και τα, Ευρωπα... και τα κοινοβούλια θα έχουν την ευθύνη για τέτοιε πράξει. Δεν μπορούμε λοιπόν να αφήνουμε όλα αυτά τα πράγματα σε ε, επιμέρου κράτη-μέλη. Τέταρτον, χωρίς κάποιο συντονισμό, τα κράτη, μέλη, τα κοινοβούλια τους μπορεί να αναγκαστούν ε, να δεχθούν κάποιες αποφάσεις τις οποίες θα αντιτίθενταν. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το είπε και ο Χάνς, ότι μπορεί κάποια κράτη-μέλη να θεωρήσουν ότι πλήττεται η φήμη τους, ότι μπορεί να μην τους βλέπουν ως αξιόπιστους εταίρους, αν δεν συμμετέχουν σε μια συγκεκριμένη αποστολή ασφαλείας. Ακόμα και δυνατά κράτη-μέλη. Ακόμη και δυνατοί ε, θεσμοί εντός κάποιων κράτων μελών μπορεί να μην τολμήσουν να φέρουν ένσταση σε κάποιες αποφάσεις που έχουν συντονιστεί ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορεί να θεωρήσουν ότι πρέπει να διατηρηθεί η φήμη τους ως συνεργαζόμενου κράτους. Ε, μπορεί να αισθανθούν ότι ε, ρηψοκινδυνεύουν θέματα αμοιβαιότητας, ότι αν αυτοί δεν συμμετέχουν, άλλοι ε, δεν θα συμμετέχουν τα αυτοί όταν έρθει η σειρά τους. Ε, σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν τα ίδια δυσκολίε στο μέλλον. Αυτό πιστεύω είναι άλλο ένα λόγο για τον οποίο θα πρέπει να υπάρχει συντονισμό μεταξύ των κοινοβουλίων. με την κατεύθυνση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάποιο βαθμό και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό, ε, αν δούμε το πέμπτο σημείο που ήθελα να τονίσω, η συνεργασία μεταξύ κοινοβουλίων, Εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπιστεί η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα κοινοβούλια ε, όταν ε, καλούν εκτελεστικά σώματα ή κυβερνήσεις πρώτων ευθυνών τους. Αυτό ονομάζεται ασύμετρη πληροφόρηση. ακούγεται πλοκό, αλλά είναι απλό. Τι σημαίνει ότι οι κυβερνήσει συνήθω γνωρίζουν περισσότερα για τα προβλήματα ασφαλεία από ότι τα, ε, τα κοινοβούλια. Πώ υπερπηδούν λοιπόν τα κοινοβούλια αυτό το πρόβλημα τη ασυμμετρία, ε, τη σύμμετρη πληροφόρηση. Ο καλύτερο τρόπο με τον οποίο τα κοινοβούλια μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα είναι αποκτώντα εμπειρογνωμοσύνη μέσα στο χρόνο. Και εδώ έχουμε το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα εθνικά κοινοβούλια. Ο χρόνος που αφιερώνουν τα εθνικά κοινοβούλια ελέγχοντας τις δικές τους κυβερνήσεις και το πώς ε, ε, συμμετέχουν αυτές σε ευρωπαϊκές ε, αποφάσεις και πολιτικές είναι χρόνος τον οποίο δεν μπορούν να αφιερώσουν στο να εξετάσουν τι κάνουν τα εθνικά κοινοβούλια σε εθνικά ζητήματα πολιτικά. Οπότε έχει νόημα να υπάρχει ένα ερετό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο θα ασχολείται πλήρως με το θέμα αυτό, το οποίο θα ειδικεύεται σε ζητήματα τέτοια και σε αποφάσεις τέτοιες και πολιτικές που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μετά οι πληροφορίες που έχει στα χέρια του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που αποκτά ε, προσπαθώντας να αποτελέσει μια γέφυρα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τα ίδια τα εθνικά κοινοβούλια κατά την επίκριση και την εξέταση των δικών του κυβερνήσεων. Η ισχυρή λοιπόν λογοδοσία των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, εξαρτάται από ένα ισχυρό Ευρωκοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Thank you. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα αρχίζει η συζήτηση. Field for, for debate, uh, Q&A. Ερωτήσεις και απαντήσεις. Πριν δώσω το λόγο σε ε, κάποιους βουλευτές. Θέλω να μιλήσω κι εγώ ως μέλος της υποεπιτροπής, όχι ως πρόεδρος. And first to, to, to Έχω μια ερώτηση στο δόκτωρα Hans Born ε, σχετικά με τη συμμετοχή της δικής μας επιτροπής ή των διαφόρων επιτροπών που θα ελέγχουν την ε, ΕΠΑ, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Έχουμε την ΚΕΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ε, Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας. Και έχουμε και την ΕΠΑ, Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Και στους δύο τομείς, ιδιαίτερα στην ΕΠΑ, οι βασικές εξουσίες είναι ακόμα στα χέρια των κρατών μελών. Uh, Έχουμε εδώ την υποεπιτροπή μας που συνδέεται με αυτό. Είμαστε υπό επιτροπή της Επιτροπής Εξωτερικών, ΑΦΕΤ, αλλά συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους, ε, γιατί συζητούμε ε, ζητήματα ασφαλείας και προβλήματα. αυτό είναι σημαντικό και για μας, και κατά την άποψή μου, είναι σημαντικό να τα συζητάμε αυτά τα θέματα. Το βάθος και το ρυθμό ε, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Αναφερθήκατε στις προκλήσεις νοτίως ε, της Ευρώπης αλλά και προς Ανατολάς. Το πρόβλημα είναι ότι η αντίληψη για τις απειλές αυτή τη στιγμή δεν είναι η ίδια παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολύ καλύτερα, μετά την παρούσα θητεία, είμαστε πιο κοντά σε μια κοινή αντίληψη για ε, τις ε, απειλές και τη δυνατότητα ή τη βούληση να εμπλακούμε σε μια σειρά τομέων και περιοχών στα πλαίσια της ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Ευρώπη δεν έχουμε τέτοια αποστολή και υπάρχει και απροθυμία γενικά. Μπορούμε να συζητήσουμε τους λόγους αν θέλετε. Αλλά είναι γεγονός. Δεν είναι ίσες όλες ε, ε, συντεταγμένες όλα τα σημεία του ορίζοντα. Και έχω την αίσθηση και τη γνώση μάλιστα ότι θεωρείται ότι αυτή η αδιαφορία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια είναι, πώς να το πω, μια συζήτηση που αφορά τα μέσα ενημέρωσης και όχι κάτι το υπαρκτό. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι παρούσες σε ευρωπαϊκό έδαφος ε, και ε, συμμετέχουν και οικονομικά. Δηλαδή δεν είναι ότι αδιαφορούν οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, και πολύ περισσότερο ε, εμείς ε, χρειαζόμαστε τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι πολιτικές μας θα πρέπει να παραμείνουν διατλαντικές. Θα πρέπει να είμαι και εγώ ειλικρινής και να σας πω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι ε, σκέφτονται την αναβάθμιση της δικής μας υποεπιτροπής σε επιτροπή. κατά την εμπειρία μου, μπορεί ε, να περιορίσει το πεδίο ενδιαφέροντος της Επιτροπής μας, γιατί στα Εθνικά Κοινοβούλια επιτροπές εξωτερικών ασχολούνται με θέματα εξωτερικών και ασφάλειας και μετά έχουμε τις επιτροπές αμήνης που ασχολούνται κυρίως με τον έλεγχο των αμυντικών ε, πολιτικών και των επιχειρήσεων των στρατιωτικών και γενικά το, την κατάσταση των στρατευμάτων. Και ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αυτά όλα είναι κάπως μετέωρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μούντι έχει το λόγο, αντιπρόεδρος της Υποεπιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους ομιλητές μας. Δεν ξέρω αν μπορώ να βάλω σε μία ερώτηση ε, ένα σχόλιο βασικά θέλω να κάνω. Δείτε με ποιο τρόπο θέλετε να απαντήσετε, αν το θεωρήσετε και ερώτηση. Ε, έχετε το δίκιο ότι έχουμε μια ε, σκληρή εξουσία για τον τρόπο που λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το έχουμε δει. Όχι αποκλειστικά από τη δική μας Επιτροπή, αλλά και με ε, το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο με θέματα δημοσιονομικά και άλλους τομείς όπου είχαμε την ευκαιρία ε, να διαδραματίσουμε το λειτουργικό μας ρόλο υπό την έννοια αυτή την νομοθετική. Αλλά αυτό θα χρειαστεί περαιτέρω εξέλιξη, διότι δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα ε, δούμε ένα ισχυρό προσανατολισμό προς την άμυνα, ε, ξεχωριστό. Εγώ έχω λίγο διαφορετική άποψη, γιατί πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια κανονική, τακτική Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας για να έχουμε αυτό το δημοκρατικό αντίβαρο απέναντι στην εκτελεστική εξουσία για να ελέγχουμε τα θέματα ασφαλείας και άμυνας as well as Και ως ε, νομοθέτης αλλά και ε, ως ε, φορέας συναπόφασης, γιατί έχει ρόλο συναπόφαση στο Κοινοβούλιο. Επομένως, το θέμα δεν είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο θα διευρύνει το πεδίο της στον τομέα αυτό, αλλά και οι ίδιες οι πραγματικότητες το επιβάλλουν στο μέλλον. More ε, Όλο και περισσότερο θα πρέπει να ασχολούμαστε ε, με τα θέματα για να τα λύνουμε, για να δρούμε σε συλλογικό επίπεδο, διότι τα κράτη-μέλη δεν θα μπορούν από μόνα τους ε, ξεχωριστά να απαντούν στις προκλήσεις που μας περιμένουν. Και έρχομαι σε ένα άλλο σημείο που αναφέρατε και οι τρεις σας και ο καθηγητής Λόρντ σίγουρα, αλλά και οι προηγούμενοι, και αυτό έχει να κάνει με τη σημασία των αξιών και των κανόνων που ε, φέρουμε σε αυτή τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δηλαδή, όχι μόνο για τις ενδεχόμενες μελλοντικές δράσεις, αλλά και για να εξισορροπήσουμε αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχομαι πάλι στο θέμα της φήμης που αναφέρατε κι εσεί και το κύριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε τι κάνει στον ανθρωπιστικό τομέα. Κοιτάξτε τι κάνει η Ένωση στη δημιουργία δυνατοτήτων και ικανοτήτων. Αλλά, ε, δηλαδή ότι συμμετέχουμε περισσότερο και σε αποστολέ. Και στο μέλλον θα πρέπει να δούμε πώς θα συγκεραστούν όλα αυτά, πώς θα εξισορροπηθούν. Εμείς παίρνουμε σοβαρά υπόψη αυτό το ρόλο. Άρα θα πρέπει να μεταξελιχθεί και αυτή η πτυχή. Όσο για τις μελλοντικές προκλήσεις, έχουμε τις νέες τεχνολογίες και το πιο δημοφιλές που συζητούν ε, πολύ είναι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στην άμυνα στο μέλλον. Γιατί αυτό συμβαίνει ήδη ανά τον κόσμο. Με ποιο τρόπο λοιπόν θα το αντιμετωπίσουμε εμείς από πλευράς κανόνων. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια τεράστια ισχύ. Αν κοιτάξετε ας πούμε κάτι που είπε χθες πολύ εύγλωτα κάποιο σε μια άλλη συνεδρίαση. Αν δείτε τις ψηφιακές πλατφόρμες που αναπτύσσονται στην Αμερική, και πώς ρυθμίζονται όλα αυτά. Η ρύθμιση είναι κάτι στο οποίο ηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει πολύ σοβαρά υπόψη να τα λάβουμε όλα αυτά. Δηλαδή βάζουμε αρχές, αξίες, κανόνες, πρότυπα. Παντού καθορίζουμε το πεδίο, αλλά και κάτι που αναφέρατε και εσείς καθηγητά Λόρντ και είναι πολύ σημαντικό και απέχουμε πάρα πολύ από τη σωστή ε, λύση. Και αυτή είναι η ε, πραγματογνωμοσύνη που έχουμε εδώ στην Ευρώπη. Και εδώ και στο κοινό. Η δουλειά μας είναι, θα μου πείτε, να είμαστε εμπειρογνώμονες. Ε, αλλά πώς θα μεταφραστεί αυτή, πώς θα μεταλαμπαδευτεί σε ένα κόσμο που λειτουργεί. Ε, όσα διαμορφώνουμε δημοκρατικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εθνικά σε ένα δημοκρατικό επίπεδο, σε εθνικά κοινοβούλια. Καταλαβαίνετε ότι είμαι από τη Βρετανία, οπότε ζω σε μια χώρα όπου έχει αποτύχει ικτρά η κοινοβουλευτική δημοκρατία και θα είμαστε εμείς παράδειγμα προς αποφυγή μάλλον και το πειραματώζω για το τι δεν πρέπει να κάνουμε για το πώς θα πρέπει να διορθώσουμε αυτή ε, τη σύνδεση ευρωπαϊκού επίπεδου και επίπεδου κράτους μέλους. Και επανέρχομαι στο θέμα της ήπιας δύναμης που αναφέρατε εσείς κύριε ε, Ράουμπε, ότι είναι πολύ σημαντικό να επεμβαίνουμε νωρίς. Αυτό το θέμα της ήπιας δύναμης επαναλαμβάνω. Και ως Βρετανοί το λέω και αυτό. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 ε, στις διαπραγματεύσεις ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας με το Κοινοβούλιο. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και άλλα πιο χρήσιμα και επικοδομητικά παραδείγματα για το πώς συμμετέχει κανείς σε πρώιμο στάδιο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μπορεί να σας ενδιαφέρει. πριν φτάσουμε να είμαστε σε μια απόφαση άσπρο μαύρο ναι όχι ή ε, απλώς επικύρωση τυπική. Πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις πάνω. Ευχαριστώ. Η κυρία Λόζινγκ. Θα μιλήσω γερμανικά. Περιμένω σύντομα να βάλετε τα ακουστικά σας. Ε, ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά πάρα πολύ περίπλοκα αυτά που μας είπατε, παρουσιάσεις και εξηγήσεις σας. Σε πάρα πολλούς τομείς συμφωνώ μαζί σας. Σήμερα έχουμε τη τελευταία μας συνεδρίαση στην παρούσα θητεία. Δέκα χρόνια τώρα συμμετέχω στην υποεπιτροπή αυτή και μέσα σε αυτά τα, τα δέκα χρόνια ο τομέας της αμυντικής πολιτικής έχει ε, ε, ε, αναπτυχθεί ραγδαία με τεράστιες ρυθμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί ε, το ενδιαφέρον της κοινή γνώμη να μην έχει εξελιχθεί αναλόγως ε, και εδώ είναι το θέμα του <laughs> αιτίου και του αιτιατού και το τι αποτέλεσμα έχει μια αιτία και ποια είναι τα ελλείμματα ενδεχομένως στην κοινοβουλευτική συμμετοχή και στις κοινοβουλευτικές δυνατότητες να έχει ένα ηγετικό ρόλο. Ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε γιατί δεν γίνονται τόσες πολλές συζητήσεις, δεν γίνει γνώμη. Έχει αναπτυχθεί πολύ ο κύριος Γιονκέρ ε, αυθολογή και ε, λέει πόσα πετύχαμε την τελευταία διετία ως προς τη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όσα πετύχαμε τα δύο τελευταία χρόνια δεν τα πετύχαμε τα τελευταία 20 χρόνια. Άρα όλο και πιο σαφές ε, είναι ότι αντίστοιχα και μάλιστα με μεγεωμετρική πρόοδο θα πρέπει να αυξάνεται και ο ρόλος ε, των κοινοβουλίων και της κοινοβουλευτικής συναπόφασης και του ελέγχου. Όποια γνώμη και αν έχει ο καθένας για τη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης. Αναφερθήκατε σε πάρα πολλά θέματα και θεωρώ πολύ σημαντικό ε, αυτό το θέμα εκ των προτέρων και εκ των υστέρων. Τώρα εμείς είμαστε εκ των υστέρων που ερχόμαστε και μαθαίνουμε τι έγινε. Καλά, αυτό χρειά μπροστά σε αυτό που θα θεωρούσε κανείς κανονικό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ε, θέλω να αναφέρω το εξής. Οι κοινοβουλευτικές δυνατότητες που έχουμε εμείς εδώ ως ευρωβουλευτές, επαναλαμβάνω ανεξαρτήτως της άποψης του καθενός, ε, ποιες είναι οι διαρθρωτικές δυνατότητες που έχουμε. Αυτό έχει να κάνει ε, και με τις πληροφορίες οποίες διαθέτουμε ως ευρωβουλευτές. Και αυτό ε, είναι πάρα πολύ δυσανάλογο μέρη. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο από εσά το είπε, ότι κανονικά εμείς θα πρέπει να είμαστε εκείνοι που θα ενημερώνουμε τα εθνικά κοινοβούλια για τον τομέα αυτό. Πάντως, ε, γεγονό είναι ότι η αλήθεια συμβαίνει ε, αντίστροφα. Όταν χρειάζομαι εγώ διάφορε πληροφορίε πιο λεπτομερεί και εμπεριστατωμένε, πρέπει να απευθυνθώ στου συναδέλφου μου στη Γερμανική Βουλή διότι εκείνοι για πάρα πολλούς τομείς γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα και έχουν πρόσβαση ό,τι έχει να κάνει ε, με το χαρακτηρισμό της διαβάθμισης λιμιτέ, περιορισμένη πρόσβαση. Ε, εμείς δεν έχουμε καθόλου πρόσβαση σε αυτή. Ε, όταν κάνουν ερωτήσεις οι πολιτικές ομάδες από τη Γερμανική Βουλή, τους απαντάνε σχεδόν αμέσως και με πολυσέλιδες απαντήσεις και εμείς δεν μπορούμε σε ερωτήσεις μας να ξεπεράσουμε 200 χαρακτήρες και το πολύ τρεις ερωτήσεις και αν είμαστε τυχεροί θα μας απαντήσουν μετά από 1,5 μήνα. Και σας ερωτώ λοιπόν, τι, πώς το βλέπετε αυτό. Τώρα μπορεί να είναι λεπτομέρεια η ερώτηση αυτή ε, σε, αυτό το περίπλοκο πλαίσιο. Πόσο καιρό θα πρέπει να περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει και να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Ε, και να συμπληρώσω κάτι. Δεν θυμάμαι ποιο το είπε. Ο κύριο Μπόρν, νομίζω. Μιλήσατε για ε, στρατό και αστυνομία. Δηλαδή έχουμε στρατιωτικές αποστολές, ε, και σε άλλα κοινοβούλια τα συζητούν, αλλά όχι τι αστυνομικέ αποστολέ. Ε, μα στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλέ αποστολέ χαρακτηρίζονται πολιτικέ, δηλαδή μη στρατιωτικέ. Και ουσιαστικά είναι αστυνομικέ, ακόμα και αν τι λένε πολιτικέ και έχουν και ένα χαρακτήρα παραστρατιωτικό. Γι' αυτό έρχεται να υπογραμμίσει πόσο σημαντικό είναι αυτά τα πράγματα να τα συζητούμε και να τα εξετάζουμε από κοινού. Μετά για τη συζήτηση αν θα είμαστε υποεπιτροπή ή κανονική επιτροπή. Αλλά εγώ δεν θέλω να αναμειχθώ σε αυτό τώρα τόσο πολύ. Απλώς να σημειώσω κάτι. Η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια με τη δημιουργία της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης έχει διευρυνθεί, επιπλακεί. Δεν έχουμε ξεχωριστούς τομεί, δεν έχουμε εξωτερική πολιτική, πολιτικά θέματα, δεν έχουμε αμυγή αναπτυξιακή πολιτική. Παντού υπάρχουν τώρα ξαφνικά ε, ε, και στρατιωτικά σκέλη. Όταν έχουμε λοιπόν μια τέτοια επιτροπή, τι θα γίνει, για παράδειγμα, όταν ε, χρήματα από την αναπτυξιακή βοήθεια πηγαίνουν σε στρατιωτικούς σκοπούς και θεωρούνται αναπτυξιακοί πόροι και έτσι ε, λογιστικά υπολογίζονται, που για μένα είναι τελείως απαράδεκτο. Ε, και ποια επιτροπή θα το συζητάει αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο για μένα αυτό και έρχεται να περιπλέξει πολύ περισσότερο τον έλεγχο, τον κοινοβουλευτικό. Μετά, τα μεμονωμένα κράτη ε, και τους διάφορους που εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Αυτό μπορούμε να το δούμε και αντίστροφα. Ας πούμε, σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Εξωτερικών, ΑΦΕΤ, συζητούσαμε για τη, διαρθρωμένη συνεργασία, τη μόνιμη, να έχουμε λήψη απόφαση κατά πλειοψηφία. Απ' τη μια λέτε ότι υπάρχουν χώρες που εκμεταλλεύονται καταστάσεις χωρίς να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Αλλά από την άλλη δεν ναι, επιτρέπεται να διαφωνούν κάποιες χώρες αν δεν θέλουν να έχουν σχέση με αυτά. Δηλαδή, ακόμα και αν οι χώρες διαφωνούν θεωρητικά, ας πούμε, με μία επέμβαση, θα πρέπει να συμμετέχουν, ε, γιατί ε, δεν είναι συνενετικές οι αποφάσεις, αλλά θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Και υπάρχουν πολύ εύθραυστα ε, οικονομικά κράτη-μέλη και άλλα πιο εύρωστα. Τώρα τι θα γίνει. Μπορεί να αποδειχθεί η κατάσταση πολύ δύσκολη για ορισμένα κράτη-μέλη. Και ένα τελευταίο. Τα εσωτερικά ζητήματα, διότι και αυτό ακούστηκε. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο τομέα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ε, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, κάτι για την πυροσβεστική ή για ε, αντιμετώπιση θεομηνιών. Υπάρχουν και ανθρωπογενείς ε, καταστροφές που δεν είναι θεομηνίες. Ε, μια γενική απεργία, ας πούμε, μπορεί σε ένα κράτος μέλος θεωρητικά να χαρακτηριστεί ανθρωπογενής καταστροφή. Και έτσι σκέφτηκαν ένα τέτοιο σενάριο. Μνημόνιο, Ελλάδα, η Γερμανία, ο ρόλος στο Συμβούλιο και τώρα Γαλλία-Γερμανία στο Συμβούλιο για τα στρατιωτικά ζητήματα και βγαίνει ο πληθυσμός σε ένα κράτος μέλος και λέει δεν τα θέλουμε εμείς αυτά τα πράγματα και αντιστέκεται. Εκεί ενδεχομένω μπορεί να κατεβάσουν το στρατό απέναντι σε αυτή την αντίσταση. Πολύ θεωρητικά τα λέω και υπερβάλλω συνειδητά για να σας δείξω πόσο ευαίσθητη είναι αυτή η συζήτηση. Γιατί και εμείς έχουμε σαφείς ρυθμίσεις για το πώς χρησιμοποιεί το στρατό στη Γερμανία. Η πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια. Ναι, ναι, τελειώνω, τελειώνω. Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί τομεί. Και τώρα με έκανε καλή πρόεδρο στην τάξη ε, και θα περιορίσω τα όσα είχα να πω. τι έλεγα. Ότι είναι πολύ ευρύ το πεδίο. Και ένα τελευταίο. Είπε η κυρία Μούντι ότι με το αμυντικό ταμείο τώρα συμμετέχουμε πολύ. Θέλω λίγο να το σχετικοποιήσω. Εντάξει, έχουμε την ευκαιρία να πούμε ναι ή όχι την άλλη φορά στις ψηφοφορίες. Με, την, την περασμένη φορά. Μετά δεν θα έχουμε ε, καμία δυνατότητα και εκ των υστέρων μπορούμε να έρθουμε να πούμε όταν αποδίδουν λογαριασμούς ότι δεν πήγανε και πολύ καλά τα πράγματα. Ευχαριστώ κυρία Βαλέρο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Είχα συγγνώμη που Άργησα να έρθω, αλλά ήμουν σε μια ψηφοφορία σε άλλη επιτροπή και έτσι λοιπόν έχασα την αρχή της συζήτησης. Μιλήσατε για την Σουηδία, από όπου και κατάγομαι, ε, και επιθεωρώ ότι είναι πολύ καλό σύστημα που έχουμε. Ε, έχουμε ένα νόμο αρχικά όταν είναι να αποστείλουμε στρατεύματα. Έτσι γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει, θα χρονοδιαγράμματα, ποια θα είναι η συμπεριφορά κτλ. κτλ. Όταν έχουμε μια πρόταση λοιπόν από την κυβέρνηση, εμείς μπορεί να την ψηφίσουμε και στην συνέχεια έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Αφγανιστάν το κάναμε αυτό ετησίως. Κάθε Δεκέμβριο λοιπόν ε, ψηφίζαμε νέα νομοθεσία για το Αφγανιστάν, διότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να το ψηφίσει, να αποφασίσει και στη συνέχεια εμείς θα πρέπει να πούμε τι είναι αυτό το οποίο κάνουν εκεί πέρα. Ασχέτως της αλυσίδας εντολής ε, θα πρέπει να ξέρουμε τι κάνουν τα στρατεύματα και να θέσουμε τους δικούς μας κανόνες. Είναι ένα πολύ καλό σύστημα. Δεν είναι χρονοβόρο. Μερικές φορές ναι, ίσως, όμως έχουμε αποστείλει στρατεύματα και πολύ γρήγορα όποτε υπήρξε η ανάγκη για κάτι τέτοιο. Οπότε και ψηφίσαμε νομοθεσίες εξίσου γρήγορα. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε τι σκέφτεστε πάνω σε αυτό. Διότι ένιωσα ότι ε, το θεωρείται πολύ χρονοβόρο, όμως είναι πολύ σημαντικό για τον έλεγχο ε, που ασκεί του Κοινοβούλιο. Και επίσης ήθελα να αναφέρω κάτι παρεμφερές με αυτό το οποίο είπε μόλις η Ζαμπίνε. Κύριε Λόγιου είπατε ότι θα πρέπει να έχουμε έναν κάποιο κοινοβουλευτικό έλεγχο σχετικά με το τι έχουμε αποφασίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, έχουμε πολλά πράγματα τα οποία εξελίσσονται και γίνονται πάνω σε θέματα άμυνας, όπως είναι για παράδειγμα το Ταμείο Άμυνα. Έχουμε το πρόγραμμα βιομηχανική ανάπτυξης, έχουμε... Ε, 30 δις αυτή τη στιγμή για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ε, και τα δύο προβλέπονται από τη συνθήκη και φυσικά εμείς έχουμε τον έλεγχο και θα πρέπει να έχουμε επίσης και τον έλεγχο να αποφασίζουμε τι θα υπάρχει στο πρόγραμμα εργασίας και τι δεν θα περιλαμβάνεται σε αυτό. Θα πρέπει να έχουμε μία άποψη πάνω σε αυτό. Όμως ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία δυνατότητα ανησυχηρίας, δεν έχουμε εκτελεστικές πράξεις, ε, οπότε Ποιο ακριβώ είναι ο έλεγχο που ασκούμε σε αυτήν την περίπτωση. Πώς βλέπετε την κατάσταση για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο όσον αφορά το αμυντικό ταμείο. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς θα μπορούμε να ασκούμε έλεγχο πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Φρόιντ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ συγγνώμη που καθυστέρησα να έρθω σε αυτή την συνάντηση είναι δύσκολο να το πιστέψουμε, όμως ένα από τα λίγα ε, από ένας από τους λίγους ευρωβουλευτές που είναι από ουδέτερες χώρες, Σουηδία και Αυστρία, δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο ότι μεγάλωσα σε αυτό το καθεστώς ουδετερότητας, όμως προσωπικά δεν ενθουσιάζομαι ιδιαίτερως με αυτή τη συζήτηση που γίνεται σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική ε, από τότε που ήρθα σε αυτό το κοινοβούλιο, πρόσφατα σχετικά, τα τελευταία πέντε χρόνια λοιπόν, αναρωτιέμαι, αρχικά χρειαζόμαστε μια ισχυρή κοινή εξωτερική πολιτική και στη συνέχεια θα μπορούσαμε να καταφύγουμε και σε μια κοινή αμυντική πολιτική. Διότι κατά τη γνώμη μου η ευρωπαϊκή δύναμη ήταν να παρεμβαίνουμε διπλωματικά. Και το τελευταίο καλό παράδειγμα είναι η συμφωνία ε, με το Ιράν για τα πυρηνικά, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν την ευρωπαϊκή στρατηγική άμυνας επειδή δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Οπότε ας προσπαθήσουμε κάτι διαφορετικό. Και δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι το θετικό. Θα πρέπει λοιπόν να συγκεντρωθούμε, να συγκεντρώσουμε όλες μας τις δυνάμεις πάνω σε μια κοινή εξωτερική πολιτική που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι ε, μια ε, πολιτική ε, που θα αφορά 500 εκατομμύρια ανθρώπους με βάση την οικονομική δύναμη που έχουμε και να μην επικεντρωνόμαστε τόσο πολύ σε κάτι το οποίο εν τέλει ίσως και να μην υλοποιηθεί. Μην με παρεξηγήσετε, δεν είμαι ειρηνιστής, δεν είμαι κάποιος ο οποίος θα πει ότι δεν θέλω καμία σχέση με τον ε, στρατό. Όμως βλέποντας την παρούσα κατάσταση, Ρωσία, Κίνα, ακόμα και οι διατλαντικές σχέσεις, οι θα πρέ... οι Ευρωπαίοι θα πρέπει κάτι να κάνουν. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουν συνέχεια τους ε, Αμερικανούς. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο όπου ε, θα χρειαζόμαστε μία λύση και στη συνέχεια ε, εμφανίζονται οι Αμερικανοί και μας βοηθάνε. Θα ήθελα λοιπόν να με βοηθήσετε ε, σχετικά με το αν ακολουθούμε τα σωστά βήματα όσον αφορά την αμυντική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η τελευταία παρέμβαση. Και τώρα θα ήθελα να δώσω τον ε, λόγο ε, στους ομιλητές μας για πέντε λεπτά στον καθένα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για όλες σας τις ερωτήσεις, σχόλια, σκέψεις. Σίγουρα θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και να εργαστούμε πάνω σε αυτά, όμως ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες από τις ε, ιδέες ε, που ακούστηκαν όσον αφορά το ερώτημα των αρχών και αξιών. ένας ε, συνάδελφος, ο Σάιμον Τζιούκ, ο οποίος ε, απεβίωσε πρόσφατα, ασχολήθηκε με το ζήτημα της πολιτικής άμυνας ε, στην έρευνά του και όταν εξέταζε τα κοινοβούλια όπου συμμετείχε και ο καθηγητής Λόρτ σε ένα πρόγραμμα ονόματι Πάκο κατέληξε λοιπόν στα συμπεράσματά του ότι ο πραγματισμός ε, μπορεί να ερμηνευθεί διαφορετικά σε αυτή την παγκόσμια στρατηγική. Όμως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το σκεφτούμε έτσι, και τα κοινοβούλια γενικότερα μπορεί να είναι οι θεσμοί οι οποίοι θέτουν τις αρχές και στη συνέχεια έχουμε τον πραγματισμό ο οποίος θα υπάρχει για την εκτελεστική εξουσία. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο είναι ενδιαφέρον και αντικατοπτρίζει τα όσα είπε ο καθηγητής, ο καθηγητής Λόρτ. Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσονται από κοινού, αναπτύσσουν από κοινού μια κοινή εξωτερική πολιτική. Και σε αυτό το πλαίσιο η θέση του Κοινοβουλίου είναι δύσκολη μαζί με τις επιτροπές από τη μία αναπτύσσετε τις, τις πολιτικές, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να τις ελέγχετε κιόλα. Το, ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας είναι ένα τέτοιο καλό παράδειγμα. Όταν το Κοινοβούλιο ε, το κοινοβούλιο συμμετείχε σε αυτό, όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να το ελέγχει κιόλα. Πώς λοιπόν μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Και μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο μέσω του ελέγχου να τηρηθούν αυτές οι αξίες. Αυτά λοιπόν έχουν αναφερθεί. Για μένα η στρατηγική άμυνας και το Ταμείο Άμυνας αρχής εξ αρχής μου φάνηκαν πολιτικά προγράμματα προγράμματα τα οποία ήθελαν να δείξουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά μπορεί να συνεργαστεί πάνω σε αυτού του τομεί, να κάνει το επόμενο βήμα της ολοκλήρωσης. Όμως και πάλι το Κοινοβούλιο βρίσκεται σε δύσκολη θέση, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, διότι υποστήριξε αυτή την ολοκλήρωση και την ε, ολοκλήρωση της ε, ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Το ερώτημα λοιπόν μακροπρόθεσμα θα είναι μπορεί να δείξει την απαραίτητη αυστηρότητα σχετικά με τις κατευθύνσεις και την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής όταν δεν θέλει να ακολουθήσει κάποιες κατευθύνσεις. Και εδώ λοιπόν είναι σημαντικό να σκεφτούμε τις εναλλακτικέ τους, πιο ήπιους τρόπους παρέμβασης. Αναφερθήκατε σε αυτό. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το ισχυρότερο όσον αφορά ε, την, τον έλεγχο και την επίβλεψη ε, των ε, ε, οικονομικών εργαλείων αλλά και των αποστολών. Έτσι λοιπόν μέσω αυτού του ελέγχου των οικονομικών εργαλείων όπως είναι για παράδειγμα το εργαλείο για την ειρήνη και την ασφάλεια συνεισφέρει στην ειρήνη και την ασφάλεια αυτό. Είναι, πρόκειται για εργαλεία όπου, ε, όπου το κοινοβούλιο μπορεί να συνεργαστεί. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται μία επιτροπή η οποία μπορεί να τα συνδυάσει όλα αυτά, το οποίο θα είναι και το πιο δύσκολο. Η Ευρωπαϊκή ε, εξωτερική πολιτική, η ΕΙΕΔ, όλα αυτά είναι ε, διαχωρισμένα μεταξύ τους. Όμως τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε δει ότι όλα ακολουθούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Και έτσι έχουμε διαφοροποιημένη λήψη αποφάσεων, όμως οι πολιτικές είναι κοινέ ουσιαστικά και χρειάζεται ένα σώμα που θα το επιβλέπει αυτό. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χανσπορν. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για τις ε, πολύ εύστοχες ερωτήσεις σας. Πολλά θα μπορούσε κανείς να πει για όλα αυτά τα θέματα. Θα επισημάνω τα σημαντικότερα. Ένα θέμα, κυρία Πρόεδρε, και χαίρομαι που το υπογραμμίσατε, δεν είναι απλά ε, οι απειλέ το ζήτημα, αλλά και το πώς τις αντιλαμβανόμαστε. Δεν είναι ένα θέμα που θα πρέπει να εκτιμούν μόνο οι επαγγελματίες στρατιωτικοί. Είναι ε, κάτι που βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων. Οπότε τέτοιες συζητήσεις πρέπει να γίνονται εδώ, στο Κοινοβούλιο και μετά να βλέπουμε πού υπάρχουν οι διαφορές. Αυτό νομίζω είναι ουσιαστικό. Το κατά πόσο μια τέτοια συζήτηση θα πρέπει να γίνεται σε επιτροπή ή σε πλήρη επιτροπή, τακτική επιτροπή, αυτοί είναι εσωτερικοί κανόνες δικοί σας. Ε, αφορούν την οργάνωση του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προσεγγίσει κανείς αυτό το ζήτημα και εσείς ε, έχετε την απόλυτη ευκαιρία να κάνετε αυτό που νομίζετε. Αλλά θεωρώ, αν ακούσετε αυτό που είπαν πολλά μέλη εδώ, ότι η σε πληρη επιτροπη τακτικη επιτροπη αυτοι ειναι εσωτερικοι κανονες δικης σας αφορουν την οργανωση του κοινοβουλιου υπαρχουν πολλοι τροποι να προσεγγισει κανει αυτο το ζητημα Ένωση επιταχύνει διαρκώς και αυξάνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και των σχετικών πολιτικών. Δεδομένου αυτού λοιπόν θα καλείται για θέματα λογοδοσίας και εξέτασης όλο και περισσότερο αυτό το κοινοβούλιο. Επίσης συμφωνώ με σας κυρία Πρόεδρε αν υπήρχε μια εξορρυκτική ε, ξεχωριστή επιτροπή θα υπάρχει πρόβλημα συντονισμού. Εάν αποφασίσετε να έχετε μια ξεχωριστή επιτροπή, οι δομέ θα είναι πολύ καλέ, οριζόντια φυσικά, με την Επιτροπή Εξωτερική Πολιτική. Όπω είπε και ο συνάδελφο από την Αυστρία, θα πρέπει να υπάρχει πολύ, πολύ καλό συντονισμό ε, τη ε, εξωτερική πολιτική με την πολιτική ασφάλεια. Επίση, ε, αυτό που συζητήθηκε για τα πρότυπα και τις αξίες ε, πιστεύω ότι είναι πολύ σωστό. Εγώ ζω στη Γενέβη, οπότε είμαι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και από έξω βλέπω ότι οι κανόνες και οι αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Όλο και περισσότερο συζητάμε ε, ποιο είναι το αφήγημα και τι υπερασπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση είναι πολύ χρήσιμη να γίνει αυτή η ενδοσκόπηση. Ε, επίσης ε, χαίρομαι που όλοι σας είδατε το σύνδεσμο των κανόνων και των αξιών ε, με την πολιτική ασφαλεία και άμυνας. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ο συνάδελφος από το Ηνωμένο Βασίλειο και ακούγοντάς σας λυπάμαι τόσο πολύ που θα φύγετε γιατί πάντα ε, συμμετέχετε επικοδομητικά στις συζητήσεις και ποιοτικά. Ε, αλλά δεν έχετε ακόμα φύγει ακριβώς, οπότε θα δούμε. Το ζήτημα της τεχνητή νοημοσύνης πιστεύω ότι θα αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία. Δύο πράγματα πρέπει να συζητηθούν εδώ. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να, να δούμε κατά πόσο πρέπει να υπερασπιστούμε την πλήρη κατάργηση τέτοιων όπλων και συζητείτε αυτό στη Γενέβη τώρα ή αλλιώς και, ή και δεν ξέρω, εσείς ως πολιτικοί θα το αποφασίσετε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο πρέπει να ζητήσουμε και το ζήτημα της σωστής, ε, της χρηστής διακυβέρνησης και λογοδοσίας ε, για αυτά τα εναλλακτικά οπλικά συστήματα και αμυντικά συστήματα. Είναι δύσκολες ερωτήσεις αυτές. Δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να δούμε τη διακυβέρνηση, γιατί αυτή η ερώτηση πολιτικά δεν είναι ορθή. Πρέπει να δούμε όμως πώς θα, τι θα κάνουμε για τα όλα αυτά ζητήματα. Μετά για το ζήτημα της Σουηδίας, ε, χαίρομαι που κάνατε αυτή την ερώτηση και εγώ το έχω επισημάνει ως καλή πρακτική. Αυτή είναι η άποψή μου. Πολύ συχνά ένα εκτελεστικό σώμα λέει τα κοινοβούλια χρειάζονται πολύ χρόνο. Αυτά είναι ανοησίες τα κοινοβουλία μπορούν να δράσουν πολύ γρήγορα αν χρειαστεί. Ε, ταχύτερα από εκεί τις κυβερνήσεις. Το εκτελεστικό λέει συχνά το κοινοβούλιο διαρρέει πληροφορίε, αλλά πολύ συχνά το αντίθετο συμβαίνει. Οι διαρροέ προέρχονται από τι κυβερνήσει πολύ συχνά. Οπότε ήθελα να, πονήσω, να τονίσω αυτή την κατάσταση, το πώ οι πρακτικέ έχουν εξελιχθεί μετά από τότε που η Σουηδία έγινε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ παλιότερα δεν είχαν αναπτυχθεί συνταγματικέ πρακτικέ σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπω είχαν αναπτυχθεί στη δική σα. Θα κλείσω εδώ να σα ξαναευχαριστήσω που με καλέσατε εδώ για να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καθηγητά Λόρτ. Έχετε το λόγο. Θα ομαδοποιήσω λίγο τις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τις τεχνολογίες, τους κανόνες, τις πληροφορίες, την εμπειρογνωμοσύνη. Το πρόβλημα είναι ότι τα κοινοβούλια ασχολούνται με, με τόσο πολύ διαφορετικά πράγματα ε, και ταυτόχρονα είναι πολιτικά ζώα διαφόρων ειδών. Αυτό το κατάλαβε ο άνθρωπος ε, ε, πριν από 170 χρόνια που είπε Καλό είναι τα κοινοβούλια να είναι χώροι συζητήσεων, να είναι λέσχες συζητήσεων και οι κυβερνήσεις να τα αποφασίσουν. Και τα κοινοβούλια θα πρέπει να έχουν ως ρόλο να εξασφαλίζουν ότι κάθε άποψη είναι αντίστοιχη με την άλλη, με επιχειρήματα. Είναι πολύ δύσκολο. Και θα πρέπει να υπάρχει ένας δημόσιος φορέας που να τα κάνει αυτά ενώπιον της κοινή γνώμης για να ε, ε, δικαιολογείται από μόνη της η κάθε άποψη. Εντάξει, αυτό είναι διαβούλευση λέγεται και θέλουμε να υπάρχει και στα κοινοβούλια. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ δύσκολο για τα κοινοβούλια να ανταποκρίνονται σε αυτό το ιδεώδες. Ένας άλλος σοφός πριν από 100 χρόνια είπε να δουλεύουν τα κοινοβούλια, να μην τρώνε όλο το χρόνο τους στην κουβέντα θα πρέπει να βοηθούν την κυβέρνηση, να τη συνοδεύουν, να την πλαισιώνουν και να παίρνουν και τις καθημερινές αποφάσεις και να εφαρμόζουν όλες αυτές τις ωραίες αρχές και τους κανόνες. Και διάφορα πράγματα που πρέπει να κάνουν τα κοινοβούλια. Λοιπόν, και να συζητούν και να εργάζονται, ε, έχουν περιορισμένο χρόνο και τα λοιπά, τα γνωστά. Και μετά θέτεται και το ζήτημα τι θα συμβεί όταν τα εκτελεστικά σώματα που προσπαθούμε να ελέγχουμε δεν έχουν ε, πολλές εξουσίες επάνω σας. Ή δεν έχετε εσείς εξουσίες επάνω τους ως κοινοβούλιο. Καλό είναι να τους συνοδεύετε και να τους πεσιώνετε, αλλά πώς τους αναγκάζετε σε ένα τομέα ε, πολιτικής. Αν δεν έχετε πολλές ε, εξουσίες νομοθετικές ή δημοσιονομικές, τι θα γίνει. Κάποιο είπε ότι δεν έχουμε δικαίωμα βέτο, κυρίας για τα προγράμματα δράσης. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι που θα μπορούσα να φανταστώ ε, για να αναγκάσετε τις κυβερνήσεις ή την εκτελεστική εξουσία, όπως και αν λέγεται, στην Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Ασφάλεια, να σας πάρουν σοβαρά έχετε το, το, την εξουσία να ε, ε, εκθέτετε και να ενοχλείτε την κυβέρνηση ε, για να ασχολούνται με θέματα που ασχολούν, απασχολούν τον τύπο και όταν οι κυβερνήσεις δεν απαντούν πιστικά μπορείτε να τις εκθέτετε και να τις τριμώχνετε. Και ένα δεύτερο, τα εκτελεστικά σώματα είναι υποχρεωμένα να σκεφτούν και το χειρότερο σενάριο. Εάν ε, πάνε τα πράγματα άσχημα για τις πολιτικές ε, και τις επικίνδυνες, όπως είναι οι αποστολές ασφαλείας, τι θα γίνει. Και κάτι που μπορεί να τους βγάλει από αυτό το χάλι, όταν τα πράγματα δεν είναι ε, καλά είναι να έχουν ακολουθήσει κάποιες διαδικασίες ε, πριν πάρουν την απόφαση και έχουν ε, δικαιολογηθεί μπροστά σε ένα κοινοβούλιο. Είπαν κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά πήγανε στραβά τα πράγματα, να πήγαμε και στο κοινοβούλιο και έγιναν όλα όπως πρέπει. Ας πούμε, προσπαθήσαμε να δικαιολογήσουμε αυτή την αποστολή πριν προχωρήσουμε και είμαστε καλυμμένοι. Και τέλος, ρωτήσατε για ε, προθύστερα σχήματα και τα λοιπά. Τι θα έρθει πρώτο και τι θα έρθει δεύτερο. Ε, η κοινή εξωτερική πολιτική ή η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Είναι εύκολο να αποφασίσεις ε, αν θα βάλεις πρώτα το κάρο ή τα άλογα, όταν είσαι, έχεις κάρο και άλογο. Όταν όμως έχεις κότα και αυγό, δεν ξέρεις αν έκανε κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Και θα πρέπει να υπάρχουν κάποια στοιχεία και όρια που μπορεί να βάζει κανείς για την εξωτερική πολιτική χωρίς πολιτική ασφάλεια. Ακόμα και αν είναι ήπια ασφάλεια ή αν είναι ε, συμμετοχή ας πούμε, στη λύση διενέξεων, συγκρούσεων και όχι την ασφάλεια με την ε, σκληρή έννοια. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Έχει λήξει ο χρόνος που είχαμε προβλέψει. Ε, σας παρακαλώ να χειροκροτήσουμε μαζί τους ε, εξαιρετικούς μας προσκεκλημένους. Colleagues, please be... Συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ για να προχωρήσουμε. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το πρόγραμμα εργασίας, το EDIDP και θα ακούσουμε τον κύριο Αλεξής, τμήματάρχη στην αρμόδια υπηρεσία όχι στην εξωτερική δράση που είπα κατά λάθο, όχι, όχι, defense ε, στη, ένα, στη Γενική Διεύθυνση Grow ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και θα μας μιλήσετε για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας. Ε, ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Bonjour, merci. ευχαριστώ και καλή σπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε ε, που μας ε, καλέσατε. Ε, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια αποτίμηση στο πρόγραμμα εργασίας του ADIDP, όπως είπατε. Αυτό έχει να κάνει με την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας. Είναι βιομηχανικό το πρόγραμμα, δεν είναι πρόγραμμα αμυντικής πολιτικής. Έχει σημασία αυτή η διαφορά ε, ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό ένας από τους βασικούς όρους είναι να συνεργάζονται τουλάχιστον τρεις εταιρείες από τρία κράτη-μέλη. Ε, ε, το ε, Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προετοιμάσει ένα πρόγραμμα εργασίας για μία διετία, αλλά οι διαγωνισμοί θα προκηρυχθούν σε αιτήσια βάση. Ο πρώτος τις επόμενες ημέρες και ένας δεύτερος στην αρχή του 2020. Το πρόγραμμα εργασίας εγκρίθηκε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 19 Μαρτίου και θα το βρείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το πρόγραμμα δράσης δεν ε, καθορίζει προφανώς έργα, project, αλλά κατηγορίες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν ε, μετά από την προκήρυξη και τον ανταγωνισμό, πώς ε, καταρτίστηκε αυτό το πρόγραμμα εργασίας. Ξεκινήσαμε από τις προτεραιότητες ε, που είχαν ορίσει οι συνομοθέτες ε, στο βασικό νομοθέτημα, δηλαδή το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όρισαν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες προτεραιότητας, προετοιμασία, προστασία, ανάπτυξη, διαχείριση της εκπαίδευσης, στράτευση και ειδικό πρόγραμμα ε, για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκεί λοιπόν βασίζεται το πρόγραμμα εργασίας. Οι δύο νομοθέτες έβαλαν τα θεμέλια και στα θεμέλια αυτά εκπονήσαμε το πρόγραμμα εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τρία βασικά στοιχεία. Το πρώτον, Όντως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις προτεραιότητες ε, αυτές που ορίζουν οι νομοθέτες στο βασικό νομοθέτημα, αλλά και μετά να αναπτύξουμε μία προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς. Δηλαδή, το αναπτυξιακό αυτό πρόγραμμα δεν αφορά αποκλειστικά κάποια κράτη-μέλη ή κάποιες μεγάλες εταιρείες, αλλά θα πρέπει να μπορεί να επιτρέπει σε όλα τα κράτη-μέλη και όλες τις εταιρείες τους να συμμετέχουν για να επιτύχει αυτό το πρόγραμμα. Το τρίτο στοιχείο, επίσης σημαντικό κατά την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας, είναι η συνοχή και η συνέπεια με άλλες δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, ιδιαίτερα ε, το CDP που είναι για τις προτεραιότητες της ικανότητες, αλλά και στα πλαίσια του ΠΕΣΚΟ, του, του μόνιμου ε, διαρθρωμένου διάλογου έτσι ώστε να συγκλίνουν στους ίδιους στόχους όλες οι προσπάθειες. Είμαστε πεπισμένοι ότι εξασφαλίζεται αυτή η συνέπεια Έχουμε κατηγορίες που συνδέονται πλήρως και συνάδουν με το CDP. Ε, σήμερα μπορούμε να υπολογίσουμε ότι περίπου 20 έργα ΠΕΣΚΟ ε, θα, από τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει αυτόματος χαρακτήρας, μετά διαγωνίζονται τα έργα, αλλά υπάρχει δυνατότητα. Ε, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο. Έχουμε ε, κάνει ε, εννέα προσκλήσεις, εκδήλωση ενδιαφέροντος το 19 και προβλέπονται 12 για το 2020 και σε αυτή τη διετία θα έχουμε δύο έργα που ονομάζονται Direct Around Direct Award με απευθείας ανάθεση, χωρίς διαγωνισμό δηλαδή στις εννέα προσκλήσεις ενδιαφέροντος έχουμε ε, όλους τους τομείς της άμυνας, ε, ξηρά, θάλασσα, ε, αέρα, ε, διάστημα και κυβέρνοχώρο. Έχουμε την επιτήρηση του αναέριου χώρου, την άμυνα στον κυβερνοχώρο επίσης και το 2019 και το 2020, πολύ σημαντικό. Επίσης έχουμε μια κατηγορία για το διάστημα, προτεραιότητα και αυτή, μια κατηγορία για την επιτήρηση στη θάλασσα, επίσης πολύ σημαντικό, ε, άλλη ε, κατηγορία για τις επόμενες ναυτικές πλατφόρμες, άλλη κατηγορία που μπορούμε να χαρακτήσουμε εγκάρσια, που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και καλύπτει εγκαρσίως διαφόρους τομείς, ε, σημαντικό αυτό για την ανάπτυξη ικανοτήτων, και άλλη ε, οριζόντια κατηγορία που έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούσε αυτό και όρο του κανονισμού. Για την κατηγορία αυτή ε, θα προκηρύξουμε δύο διαγωνισμούς, τον ένα το 2019 με 7,5 εκατομμύρια ευρώ και 10 εκατομμύρια θα ακολουθήσουν το 2020. Ε, προτείναμε να διαφοροποιήσουμε τη χρηματοδότηση στις δύο χρονιές αυτές για να προετοιμαστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει, Γιατί αυτή τη στιγμή προκυρήσεις στο διαγωνισμό έχουν πολύ γραφειοκρατία οι μικρομεσαίες για να ετοιμάσουν την υποψηφιότητά του. Όσε λοιπόν δεν μπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητα το 19 να προετοιμαστούν για το 2020. Όπως σας είπα υπάρχουν και δύο έργα που έχουν να κάνουν με την άμεση ανάθεση που προβλέπει ο κανονισμός και αναφέρονται στο πρόγραμμα αυτό. Το είναι το Euromar που είναι το νέο drone με περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ σε μία διετία. Είναι σύστημα ε, drones που δεν υπάρχει στην Ευρώπη και απαντά στα κριτήρια του κανονισμού. Και ένα δεύτερο project ε, με άμεση ανάθεση αφορά το ESOR που είναι ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ε, ασφαλής 37 ε, εκατομμύρια ευρώ ε, πάλι για τη διετία. Αυτά είναι με άμεση ανάθεση. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. Υπάρχει δυνατότητα, αλλά δεν έχει καταλήξει η απόφαση στο πρόγραμμα εργασίας ε, μόλις ολοκληρωθεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσει αυτούς τους ομίλους ότι μπορούν να το αναλάβουν άμεσα, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να φέρουν όλα τα δικαιολογητικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποδεικνύοντας ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας αφενός και αφετέρου ότι πληρούν και τα κριτήρια για την άμεση ανάθεση. Και μόνο όταν γίνει αυτή η ανάλυση και αξιολογήσουμε αν πληρούνται αυτά τα κριτήρια, οι όμιλοι θα μπορέσουν να λάβουν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το ποσό τώρα που θα δοθεί σε κάθε εταιρεία, αυτό θα εξαρτηθεί από τον τύπο δράσης που προτείνουν οι όμιλοι. Ξέρετε ότι ο κανονισμός προβλέπει 20% για τα πρωτότυπα και μέχρι και 100% για τις άλλες δράσεις. Ε, στις προκηρύξεις διαγωνισμών ε, θα αναφέρουμε ότι για τα πρωτότυπα και για τα υπόλοιπα η αρχική χρηματοδότηση είναι πιο χαμηλή. Γιατί ε, από τον κανονισμό προβλέπεται και ένα σύστημα μπόνους πρημοδότησης των μικρομεσαίων και κυρίως των διασυνοριακά λειτουργούσα και για τις δράσει από το, την ΠΕΣΚΟ, τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία. Δηλαδή, αν δίναμε από την αρχή το 100% θα χάναμε τον πόνου της πρημοδότηση για τις μικρομεσαίες. Άρα στην αρχή έχουμε 65% εκταμίευση για όλες τις δράσει, πράγμα που επιτρέπει ακριβώς να αφήσουμε ένα 35% για πρημοδότηση και να έχουμε το σύνολο 100% μετά. Για τα πρωτότυπα, εκεί το αρχικό κατόφλι είναι 20% και ενδεχομένως με μπόνους και με πρημοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι και 35%. και για τα σχέδια της μόνιμης ε, διορθωμένης συνεργασίας. Ένα άλλο σημαντικό που καμιά φορά προκαλεί σύγχυση, πρημοδότηση των μικρομεσαίων δεν αφορά ε, το πριμ μόνο για τις μικρομεσαίες, αλλά και για ομίλους που συμπεριλαμβάνουν ε, μικρομεσαίες ε, εταιρείε. Δηλαδή μπορεί να είναι μεγάλες, αλλιώς δεν θα υπάρχουν και κίνητρα. Και ένα τελευταίο στοιχείο για τα διαδικαστικά και το χρονισμό. Η προκήρυξη για το 19 θα βγαίνει όλα πάρα καλά μεθαύριο στις 4 Απριλίου και θα μπορέσουν να υποβάλουν την υποψηφιότητα της εταιρείας μέχρι τα τέλη Αυγούστου και αφού λάβουμε τις προτάσεις αυτές, ε, τις υποψηφιότητες, θα εξετάσει και θα επαληθεύσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας και στη συνέχεια τα κριτήρια για την άμεση ανάθεση με τη βοήθεια ε, ανεξάρτητων εμπειρογνωμών. Και με βάση αυτά θα καταρτήσουμε ένα κατάλογο δικαίουχων επιχειρήσεων και αυτός ο κατάλογος αναμένεται να είναι έτοιμος περί τα τέλη του έτους. Ταυτόχρονα εργαζόμαστε ε, για την προετοιμασία της προκήρυξης διαγωνισμού του 2020 που μπορεί να προκηρυχθεί ε, στις αρχές του έτους από το Γενάρη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Mm-hmm. Actually, δεν έχει ζητήσει κανένας το λόγο. Ε, κύριε Ποντή, μήπως... Ευχαριστώ πολύ. Για την ώρα. Ήταν ένα ερώτημα διευκρίνησης. Ίσως η συνάδελφος να έχει πιο αναλυτικές ερωτήσεις. μιλήσατε για τις εννέα προσκλήσεις που άνοιξαν για την περίοδο 19-20. Όμως ρώτησα ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ε, αφορά τις εταιρείες οι οποίες θα επιλεγούν ε, στο τέλος της χρονιάς ε, και αν ισχύει αυτό τότε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τις δύο προτάσεις flagship. Ε, συγγνώμη αν δεν κατάλαβα ακριβώς τις ε, λεπτομέρειες. Θα ήθελα να ξέρω ακριβώς ε, σχετικά με το πώς θα προγραμματιστεί αυτό. Και όσον αφορά το πρόγραμμα, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση προηγουμένως που ίσως να την ακούσατε όμως όσον αφορά την ενασχόληση με το Κοινοβούλιο και το να ε, συνεργάζεται περισσότερο μαζί σας πάνω σε αυτή τη διαδικασία, ε, σας ε, παρουσιάζουμε πολύ γρήγορα την... Ακούσαμε πολύ γρήγορα αυτή την πρόταση, οπότε θα ήθελα να ακούσω και άλλες προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε περισσότερο πάνω σε αυτό. Η κυρία Λούιζη Έχω μία ερώτηση σχετικά με τις ε, συνεισφορές ε, της Επιτροπής ε, θα προσθεθεί με τον παράγοντα 5 ε, για την, εθνικά, ε, για την εθνική χρηματοδότηση. Έχει συμβεί αυτό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού drone, ε, διότι εκτός από τα 100 εκατομμύρια θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα 500 εκατομμύρια από τα κράτη-μέλη. Και εδώ ποια κράτη-μέλη και πόσο έχουν πληρώσει μέχρι στιγμής ή πόσα έχουν εγκρίνει. Και το ερώτημα, επόμενο ερώτημα είναι στις 19 Μαρτίου η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ε, ποια προγράμματα θα λάβουν αυτά τα 520 εκατομμύρια. Τώρα πότε ακριβώς το Κοινοβούλιο έλαβε για πρώτη φορά αυτόν τον κατάλογο και πώς ακριβώς ε, προχώρησε η κοινοβουλευτική διαδικασία και απόφαση πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης να διευκρινίσετε περαιτέρω για την ε, μελλοντική ε, πλατφόρμα, ναυτική πλατφόρμα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα για, για τις κατηγορίες ε, για τις προκηρύξεις, ναι, ε, εννέα κατηγορίες θα προκηρυχθούν το 2009. Για το 2019 ταυτόχρονα θα προτείνουμε δύο έργα άμεσα ανάθεσης. Δεν θα συμπεριλαμβάνονται δηλαδή στα calls για τα Eurodrones και για το ESA δεν θα αποτελέσει κομμάτι αυτό των διαγωνισμών. Αυτό σημαίνει ότι στις επόμενες εβδομάδες η Κομισιόν θα γράψει στο consortium, στα consortium που στις κοινοπραξίες που ενδιαφέρονται. Θα τους ε, αναφέρεται η απόφαση της Κομισιόν όπου προβλέπεται ε, παραχώρηση χ εκατομμυρίων για την ανάπτυξη δράσεων στο πλαίσιο αυτών των έργων θα ζητήσουμε από τις κοινοπραξίες διευκρινήσεις για τα κριτήρια επιλεξιμότητας, για τις συγκεκριμένες δράσεις που μπορούν να αναπτύξουν, για την υλοποίηση όχι των κριτηρίων που θα υπάρχουν στον κανονισμό. Αυτό θα συζητηθούν τους επόμενους μήνες και μετά από την εξέταση αυτή, από τον έλεγχο του κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια, η Κομισιόν θα προτείνει να ε, δοθεί να δοθούν ποσά σε αυτή την κοινοπραξία. Είναι δύο ε, διαδικασίες λοιπόν παράλληλες. Για τη ε, call του 2019 όσον αφορά τη διαδικασία και το χρονοδιαγράμμα μετά από την παραλαβή των προσφορών πιστεύουμε ότι μέχρι τον έτος θα έχουμε αναλύσει όλες τις προτάσεις που θα έχουν επιλεγεί και συνεπώς θα πρέπει να έχουμε τον κατάλογο των, προπο... των προτάσεων που έχουν επιλεγεί για το 2019. Μετά πρέπει να συζητήσουμε τις τεχνικές διατάξεις. Οι συμφωνίες θα υπογραφούν προφανώς ε, αρχές του επόμενου έτους και για την άμεση ανάθεση. Ε, το χρονοδιάγραμμα θα είναι περίπου το ίδιο γιατί μέχρι να απαντήσουν οι κοινοπραξίες θα πρέπει να γίνει ανάλυση, να ελέγξουμε τα ζητήματα ασφαλείας. Οπότε πιστεύω θα έχουμε φτάσει Χριστούγεννα ήδη. Και για το 2019 η διαδικασία θα είναι ίδια μόνο από το 2019 θα μπορούμε να δημοσιεύσουμε τις προσκλήσεις από τον μήνα Ιανουάριο, οπότε θα είναι πιο γρήγορη για το 20. Euh, euh, euh, για τα Eurodrones προβλέπεται αυτή τη στιγμή πράγματι ένα ποσό 100 εκατομμυρίων ε, για διάστημα δύο ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρήχαν τα κράτη-μέλη στο ε, πλαίσιο της Επιτροπολογίας, στόχος ε, είναι η χρηματοδότηση μελετών σκοπιμότητας και σχεδιασμού για την ανάπτυξη των ε, εξοπλισμών αυτών. Η χρηματοδότηση αυτή δεν θα φτάσει ποτέ το 100% όπως ενδεχομένως προβλέπει ο κανονισμός γιατί για τη σκοπιμότητα και το σχεδιασμό η Κομισιόν μπορεί να πάει μέχρι το 100% του κόστους. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί, πολύ απλά διότι είναι 500 εκατομμύρια ο προπολογισμό. Αν βάζαμε 100% σημαίνει ότι θα βάζαμε 500 εκατομμύρια μόνο γι' αυτό. Αυτό είναι αδύνατον. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα είναι πολύ χαμηλότερη δαπάνη για αυτά τα έργα. Δεν έχουμε τα νούμερα αυτή τη στιγμή. Αναμένουμε τι διευκρινήσει από τα κοινοπραξίε, αλλά σίγουρα δεν θα υπερβούμε το 15-20% του πραγματικού κόστου τη δράση. Τι σημαίνει ότι αν χρηματοδοτήσουμε το 20% τότε τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν το 80%. Αυτή είναι η λογική του EDDB. Λέει ότι η Κομισιόν πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί ώστε τα κράτη-μέλη να οικειοποιηθούν τα έργο ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χαθεί η κοινωτική χρηματοδότηση αλλά ότι ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη θα θεωρούν ότι πρόκειται για μια ε, για εξοπλισμού σημαντικού, του οποίου χρειάζονται και του οποίου θα χρηματοδοτήσουν. Και στο τέλο ε, θα το αγοράσω, στο τέλο τη διαδικασία ενδεχομένω. Οπότε τα κράτη-μέλη είναι αυτά που θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν τη διαφορά. Όσον αφορά την προετοιμασία του προγράμματος εργασιών, αυτό γίνεται βάσει του κανονισμού IDDP, δηλαδή της επιτροπολογία. Γνωρίζουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και το κείμενο, εφαρμόζουμε ουσιαστικά το κείμενο ως έχει. Κατά την εκπόνηση των εγγράφων για την επιτροπολογία εστάλησαν οι πληροφορίες. Όταν κάθε η Επιτροπή Προγράμματος να συζητήσει την προετοιμασία του προγράμματος, δημιουργούμε ένα χρονοδιάγραμμα, πρακτικά, μια ημερήσια διάταξη και όλα αυτά διαβιβάζονται στα θεσμικά οργάνα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κανονικά στέλνονται όλα αυτά τα στοιχεία κατά τη φάση προετοιμασίας. that... Νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν. Ήταν πολύ ολοκληρωμένη αυτή η ενημέρωση για το πρόγραμμα εργασιών του EDIDP. Το θέμα θα μας απασχολεί διαρκώς. Ήταν ένα από τα σημαντικά ζητήματα συζήτησης εδώ στην υποεπιτροπή μας. Και υπολογίζουμε να συνεχίσει να είναι στην επόμενη θητεία. Σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ μην αποχωρήσετε, θα ξεκινήσουμε ξανά σε λίγα λεπτά. Σε πέντε λεπτά περίπου θα έρθει ένας ε, πολύ ενδιαφέρον ομιλητής για ένα πολύ ενδιαφέρον σχολείο. Colleagues, Συνάδελφοι, παρακαλώ, καθίστε. Περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης. Και ε, το τελευταίο σημείο όλης της θητείας. Θέλαμε έτσι να την στέψουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα της ε, αναδυόμενες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Ε, με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω για άλλη μια φορά τον ε, κύριο Πέντρο Σεράνο, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα στην ΕΙΕΔ, γνωστό σε εσάς φυσικά και του είμαστε ευγνώμονες που ξανά έρχεται εδώ για τη συζήτηση αυτή. Δεύτερο, αριστερά μου είναι ο κύριος ε, Γιάν Χαβρανέκ, ε, σύμβουλος πολιτικής ε, στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, γνωστός μας επίσης σε πολλούς από εμά και εξίσου σημαντικός ο εμπειρογνώμων κύριος Τόμας Βάλασεκ, διευθυντής της Carnegie Europe. Συναδελφοί, το θέμα είναι οι προκλήσεις αυτές και είναι ένα δύσκολο θέμα και ξεκινάμε τη συζήτηση. Κύριε Σεράνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαρά μου. Ε, έρχομαι στην Επιτροπή σας. Θέλω οπωσδήποτε να αποτίσω ένα φόρο τιμής στο έργο της Επιτροπής σας κατά τη διάρκεια της παρούσης κοινοβουλευτικής περίοδου και τη εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και πόσο μας ενθαρρύνατε να προχωρήσουμε σε αυτά που είναι σημαντικά βήματα ε, για να προωθήσουμε τα θέματα αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι οι προκλήσεις που μας περιμένουν. Πριν από αυτό όμως, θα ήθελα να πω το εξής. Είναι πραγματικά τρομακτικές αυτές οι προκλήσεις. Και κατά κάποιο τρόπο είναι και οι ίδιες αυτές που είχαμε πριν από μία πενταετία στην αρχή της θητείας. Ωστόσο κάτι κερδίσαμε το τελευταίο διάστημα και την τελευταία τριετία. Έχουμε περισσότερη επίγνωση για το ποιες είναι οι προκλήσεις, πώς συνδέονται μεταξύ τους, αλλά και πώς θα αποκρινόμαστε εμείς σε αυτές. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάναμε σημαντική πρόοδο και έχουμε οπλιστεί για να απαντούμε σε αυτές ε, που είναι και περίπλοκες με τρόπο πιο ενωμένο. Θα αναφερθώ λεπτομερώς στη συνέχεια. Και αυτό δεν μπορεί να το επομίζεται ε, ένα ή δύο διαφορετικά μέσα. Θα πρέπει να κινητοποιούμε όλη την ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για να επιτυγχάνουμε. Και θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω κάτι ακόμα. Το ρόλο που έπαιξε η παγκόσμια στρατηγική που παρουσίασε το 2016 η κυρία Μογκερίνη ε, μας έδωσε βασικά στοιχεία, κλειδιά για να ε, ερμηνεύουμε την πραγματικότητα στην οποία ζούμε, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και πώς ε, κινητοποιείται η απόκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι περισσότερες προσπάθειές μας ε, ακολούθησαν αυτή τη στρατηγική. Έθεσε το πλαίσιο λοιπόν η κυρία Μογκερίνη και ακολούθησαν ε, ε, με συγκεκριμένες δράσεις με βάση τις ιδέες της για την παγκόσμια στρατηγική. Ένα λοιπόν από τα βασικά ε, σημεία και απαντήσεις είναι ότι αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, θα πρέπει να προχωρήσουμε προς μια πιο ενεργή διεθνή παρουσία Βλέπουμε απειλέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να είναι η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα ή οι ε, ανεξέλεκτες μεταναστευτικές ροές. Δεν πρόκειται να τα λύσουμε αυτά εάν περιχαρακωθούμε και κλειδωθούμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να έχουμε αποτελεσματικότητα πρέπει να έχουμε πιο ενεργή διεθνή παρουσία. Αυτό είναι το βασικό. Και να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να εδρεώνει το ρόλο της ε, στο παγκόσμιο σκηνικό για να προστατεύει, να προωθεί τις αξίες και τις αρχές της αλλά και τα συμφέροντά της και αυτό λοιπόν είναι κάτι που κατανοήσαμε καλύτερα τα τελευταία χρόνια και που συνεργαζόμαστε σε αυτό και με την υποστήριξη φυσικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας. Αν δούμε λοιπόν τις ίδιες τις προκλήσεις, μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση περιβάλλεται από κρίσεις. Αυτό ίσχυε και πριν από μία πενταετία. Και δυστυχώς δεν εξαφανίστηκαν αυτές αυτό χαρακτηρίστηκε κυρίως ε, στην περίοδο ε, του 2011 και το 2014. Το 2011 ήταν η Αραβική Άνοιξη, αλλά δεν καταλαβαίναμε πολύ καλά τι συνέβαινε στον κόσμο. Και μετά τώρα το 2019 έχουμε δει τα αποτελέσματα αυτής της Αραβικής Άνοιξης με διάφορους τρόπους. Και κατανοούμε καλύτερα ποιες ήταν οι δυνάμεις πίσω από τα κινήματα αυτά και ποιες είναι οι πραγματικότητες στις οποίες σήμερα ε, αντιμετωπίζουμε και πρέπει να ξεπεράσουμε. Ως συνέπεια του 2011 θα ανέφερα κυρίως ε, τρία ε, προβλήματα ε, που μας αφορούν. Κρίση στη Μέση Ανατολή, Συρία, Ιράκ και η Εμένη. Το 2015, 14 μάλλον άρχισε αυτό, ήταν ακόμα η αρχή και το 2011 πόσο μάλλον, μετά το 2014 ήταν η μέση της κρίσης, τώρα φαίνεται να τελειώνει η κρίση στη Συρία και ο πόλεμος στο Ιράκ. Αλλά η κρίση δεν έχει ε, εξαφανιστεί. Τα θεωρούμε με μονομένες σειράξεις στη Συρία, στο Ιράκ, στην Ιεμένη. Δεν είναι ε, ξεκομμένες αυτές οι σειράξεις, εντάσσονται σε μια περιφερειακή αναζήτηση για μια νέα ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή και δεν έχει τερματιστεί αυτή η διελκυστίδα, συνεχίζεται ακόμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Και έχουμε δει μερικέ από τις συνέπειες. Έχουμε νέα μάρκα δυστυχώς τρομοκρατία στον ΤΑΕΣ, στο Ισλαμικό κράτος και άνοιξαν και δρόμοι όχι μόνο για τη μετανάστευση, αλλά πολλοί από εκείνου που το 2015 ανησύχησαν τόσο πολύ την Ευρώπη, που είχαμε περίπου ένα εκατομμύριο μετανάστες που ήρθαν, οι περισσότεροι από αυτούς, πολλοί από αυτούς προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και πρέπει να το κατανοήσουμε και έχουν ένα θεμητό αίτημα για διεθνή προστασία. Γεγονό είναι βέβαια ότι όταν ανοίξει ένα μεγάλο δρόμο θα ακολουθήσουν και θα παρισφρήσουν και πολλοί άλλοι. Πράγμα που συνέβη. Αλλά αυτέ ε, ήταν οι άμεσε συνέπειε για την ασφάλεια τη Ευρώπη. Αλλά το πρόβλημα υπερβαίνει αυτέ τι εκδηλώσει και είναι ένα ε, ε, μεγάλο περιφερειακό πόλεμο που δεν έχει λυθεί και κλείσει. Δεύτερο μεγάλο θέατρο πολέμου η Λιβύη που οδήγησε και σε κάποιο βαθμό ε, στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Εκεί ακόμα δεν έχουμε βρει λύση, παρόλο που εγκρίναμε σημαντικά μέτρα. Και αυτή η αποσταθεροποίηση στην ε, Λιβύη εξακολουθεί να μας ε, απειλεί και ξέρετε τις μεταναστευτικές ροές μέσω της Λιβύης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν σταματήσει. Και ένα τρίτο στοιχείο ε, των ε, επιπτώσεων του 2011 είναι η κατάσταση στο Σαχέλ. Από σταθεροποιήθηκε από τον πόλεμο στη Λιβύη, το είδαμε αυτό το 2012. Το Μάλι περίπου το κατέλαβαν οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες ολόκληρο και αποσταθεροποιήθηκε η περιοχή του Σαχέλ ε, που ίσως ε, έπρεπε να είμαστε πιο ενεργοί ε, με την αναπτυξιακή βοήθεια, την ανθρωπιστική, τις αποστολές της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Έχουμε παρουσία, αλλά μας ανησυχεί και ιδιαίτερα ο συντονισμός των χωρών αυτών και η συνένωσή τους έτσι ώστε να μπορέσουν να εδραιώσουν και να επιβάλλουν τη σταθερότητα στην περιοχή. ξέρετε ότι έχουν συνενωθεί πέντε χώρες του Σαχέλ στο G5. Έρχομαι τώρα στο 2014. Ε, υπάρχει και το 2008 βέβαια που ήταν το ανατολικό μας μέτωπο και η σχέση μας με τη Ρωσία και οι δράσεις που, ε, στις οποίες προέβη η Ρωσία. Είχαν έναν αντίκτυπο γιατί παραβίασε την εδαφική ακαιρεότητα της Γεωργίας τότε, το 8, και της Ουκρανίας αργότερα το 14, με την προσάρτηση της Κρυμαίας που φυσικά εμείς απορρίπτουμε ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν και άλλες ενεργές εστίες ανάφλεξης, ε, Μολδαβία, Υπερδνηστερία ή και το ορεινό Καραμπάχ. Και εδώ ο ρόλος της Ρωσίας έχει έρθει στο προσκήνιο. Ε, ανακαλύψαμε μετά ή ανακαλύψαμε ε, ξανά νέες απειλές, υβριδικές τις ονομάζουμε, με μια σημαντική διάσταση ε, στον κυβέρνοχώρο και η σχέση μας με τη Ρωσία έχει αλλάξει δραματικά την τελευταία πενταετία. Από εταίρος με τον οποίο είχαμε ε, δύο συνόδους κορυφής το χρόνο, έχει καταντήσει μια χώρα με την οποία έχουμε σημαντικές διαφορές φυσικά, ιδιαίτερα και κυρίως λόγω της παραβίασης της εδαφικής ακαιρεότητας της Ουκρανίας και της Γεωργίας. και έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ οι σχέσεις μας. Ένα τρίτο στοιχείο το οποίο θέλω να αναφέρω Το τρίτο λοιπόν αυτό στοιχείο είναι η αναγέννηση δυστυχώς γεωστρατηγικών αντιπαλωτήτων. Εδώ έχουμε την κατάσταση της Ρωσίας που σας ανέφερα προηγουμένως αλλά με πιο ενεργή συμμετοχή σε διεθνή μέτωπα, πολύ πέραν των συνόρων της. Αλλά έχουμε επίσης και μια πιο δυναμική Κίνα, έτσι, που μπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο και οικονομικά και τεχνολογικά επεκτείνεται, αλλά και γίνεται σίγουρα η δεύτερη παγκόσμια οικονομία ε, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, τρίτη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αναβαθμίζεται και ο ρόλος της στη διεθνή πολιτική. Πολύ σημαντικό. Επίσης βλέπουμε αλλαγές και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Με την πολιτική πρώτα η Αμερική, που είχε πολλές συνέπειες ε, με την μονομερή δράση σε πολλές φορές, με την αμφισβήτηση της πολυμερού συνεργασίας επανελειμμένα και σε διάφορα φόρα και σε πολλά θέματα κλειδιά ακολουθούν ε, το δικό τους μοναχικό δρόμο. Παρόλο που οι Ηνωμένε Πολιτείε παραμένουν ε, ο μεγαλύτερος ε, διεθνή εταίρο Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορικά, όλε αυτέ οι εξελίξει επηρεάζουν τη σχέση μα. Έτσι λοιπόν έχει το νέο περιβάλλον που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε γεωστρατηγική αντιπαλότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάπου θα πρέπει να βρει εκεί τη θέση της. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, μειώνεται ο πληθυσμός, ε, μειώνεται το οικονομικό βάρος, το ειδικό της ε, Ένωσης και υπάρχουν και άλλοι μακροοικονομικοί δείκτες. Παρ' όλα αυτά, ως Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουμε μίζων ε, διπλωματική, βιομηχανική, οικονομική δύναμη, ακόμα και αμυντική. Αν δείτε το σύνολο προπολογισμό, τον αμυντικό για όλα τα κράτη-μέλη, ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν παραμένουμε από τους πρώτους ή ε, από τις πρώτες υπερδυνάμεις, γιατί να μην το πω. Αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δρούμε και ως υπερδύναμη και με τις ικανότητες και τις δυνατότητες που έχουμε να μπορούμε να προάγουμε ε, τα συμφέροντά μας και να υπερασπιζόμαστε και να προασπίζουμε τις αξίες μας. Αυτό κάνουμε τώρα. Με αυτές τις απειλές και ε, σε μια κρίσιμη καμπή για να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινητοποιήσει όλη τη την ενέργεια για να αποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις. Αυτό δεν γίνεται μόνο με μέσα ασφάλειας και άμυνας. Θα πρέπει να είμαστε πιο σοφοί ε, ως προς την οικονομία, την βιομηχανία, το πώς προστατεύουμε τον κυβερνοχώρο μας, ακόμα και το διάστημα. Αλλά παίζει ρόλο ε, η άμυνα και στην Επιτροπή σας. Και τα τελευταία χρόνια συλλογικά ήμασταν πάρα πολύ δραστήριοι στην πρόθεση μέσων και εργαλείων που θα δώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη αμυντική ικανότητα. Με μέσο διάφορα συνεργασία, τα γνωρίζετε πολύ αυτά. Δεν θα μπω σε περιγραφές, πέσκο φυσικά, η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία και τα διάφορα αμυντικά ε, χρηματοδοτικά μέσα με το αμυντικό ταμείο, το, το ΚΑΡΤ, με ε, διάφορα άλλα αρχικά, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που κάναμε για την ανάπτυξη των ικανοτήτων, για τη διαχείριση των χρήσεων με πρωτοβουλίες ε, που διευρύνουν ε, τη δυνατότητά μας και για τη διαχείριση των κρίσεων με πολιτικά μέσα, μη στρατιωτικά δηλαδή, Ακόμα συζητείται ε, η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση, ο Μηχανισμός για την Ειρήνη μάλλον, ε, για την αμυντική συνεργασία, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερη συνεισφορά στην παγκόσμια ασφάλεια και ειρήνη. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στη συνεργασία με τους διαφορού εταίρου. Βεβαίως, γνωρίζουμε πάρα πολύ ότι είμαστε πρωταγωνιστές ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κανένα πρωταγωνιστής δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ε, το μέγεθος των προβλημάτων και των προκλήσεων που σας ανέφερα. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργάζεται με εταίρου. Τι να κάνουμε. Και τα τελευταία χρόνια ε, ε, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και ε, και προσοχή στη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Τον Ιούλιο του 2016 και τον Ιούλιο του 2018 είχαμε, είχαμε δύο κοινέ διακηρύξεις, 7 τομείς ε, δραστηριοτήτων με 74 κοινέ δράσεις που ουσιαστικά έχουμε δημιουργήσει μια πρακτική μόνιμη συνεργασία σε επίπεδο επιτελείων με τον ΝΑΤΟ. Τώρα διευρύνουμε και επεκτείνουμε ε, τις διάφορες δομές μας ε, σε κρατικό επίπεδο, αλλά η σχέση μας και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άμυνα ταιριάζει γάντι με τη διευρυμένη σχέση με τον ΝΑΤΟ. Και όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που σας ανέφερα για την άμυνα, για τη διαχείριση των κρίσεων θα είναι πρωτοβουλίες που θα συνεισφέρουν για να ε, έχουμε επιμερισμό των βαρών στη Διατλαντική Συμμαχία και την ανάπτυξη ικανοτήτων ε, ε, που ε, ευθυγραμμίζεται και με τις ανάγκες και με τις απαιτήσει του ΝΑΤΟ. Δηλαδή ήταν πυλώνας πραγματικά το ΝΑΤΟ σε αυτά τα θέματα τα αμυντικά και ασφαλεία τα τελευταία χρόνια. Όπως ήταν και η σχέση μας με τα Ηνωμένα Έθνη που εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ισχυρή στη διαχείριση των κρίσεων αλλά και στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και στη μη διάδοση και τον αφοπλισμό και ε, για μια τελευταία αναφορά στην Αφρική. Πολλές από τις κρίσεις που αντιμετωπίζουμε προέρχονται από την Αφρικανική Ήπειρο. Και τώρα έχουμε ένα ε, μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψαν οι δύο πρόεδροι ε, των δύο επιτροπών Ευρωπαϊκής και Αφρικανικής Επιτροπής πέρυσι. Έχουμε τακτικό διάλογο με την Αφρικανική Ένωση στον τομέα της ασφάλειας, της άμυνας και της διαχείρισης των σχετικών τους κρίσεων. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ε, ένα πιο πολυμερές πλαίσιο, πιο στιβαρό για να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και με πολύ μεγάλη χαρά να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να έχετε για αυτά τα θέματα και για άλλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεράνο. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γιάν Χάβρα Νέκ, Σύμβουλος Πολιτικής ε, από την Γενική Γραμματεία του ΝΑΤΟ. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη ε, δυνατότητα που μου δίνετε σε αυτή την τελευταία συνεδρίαση και να μιλήσουμε για τις αναμειδιόμενες ε, απειλές για την ασφάλεια. Θα ήθελα να σας μιλήσω και ως ε, ιδιωτικός πολίτης, ο οποίος νοιάζεται για την Ευρώπη και την διατλαντική συνεργασία και δεν θα περιοριστώ μονάχα στην επίσημη μου θέση ως εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων ε, πραγματικά ε, κοιτά προς το μέλλον, όμως θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία και να αναφέρω και το παρελθόν. Το 2019 ήταν μια χρονιά εορτασμών. Σε δύο μέρες ε, οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν στο ΝΑΤΟ για να γιορτάσουν την 70η επέτειο ε, την ε, διεύρυνση του ΝΑΤΟ και την προηγούμενο μήνα γιορτάσαμε και άλλες διευρύνσεις του ΝΑΤΟ Οπότε είναι σημαντικό να πούμε ότι χωρίς τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ε, ε, χώρες που μπήκαν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ήταν τόσο εύκολο να το πράξουν αυτό στο παρελθόν. Από το 2014 λοιπόν έχουμε μία άνευ προηγουμένου χειροτέρευση της συνθήκης ασφαλείας όπως περιέγραψε ο πρέσβης Σεράνο ε, το οποίο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερος από την επέμβαση της Ρωσίας ε, στην Ουκρανία ως ανταπόκριση ε, το ΝΑΤΟ έχει αναλάβει την μεγαλύτερη ενίσχυση της άμυνας της, Ευρωπαϊκής, της Ευρώπης από το 1989 και έπειτα. Αυτή η προσαρμογή έχει καταστήσει πιο εύκολη την περιοχή. Παρ' όλα αυτά ο πλανήτης παραμένει ένας επικίνδυνος κόσμος. Η Ρωσία παρα... συνεχίζει να μην τηρεί διεθνείς ε, συνθήκες, ε, αμφισβητεί και δοκιμάζει την ενότητα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνει σε κυβερνοεπιθέσεις επίσης ε, αναμειγνύεται στις δημοκρατικές διαδικασίες ε, και η Μόσχα συνεχίζει την ε, στρατιωτική της ενίσχυση στη Νότια Ευρώπη τώρα, όπως είπε ο πρέσβης Σεράνο, υπάρχει περιορισμένη πιθανότητα ειρήνης παρά την ήττα του ISIS και στο μεταξύ η Κίνα εμφανίζεται ως ένας στρατηγικός ανταγωνιστής ε, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Δημο, διπλωματία, εμπόριο, οικονομία, όλα αυτά συμβαίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό στον κυβερνοχώρο και οφείλω να ομολογήσω ερχόμενος εδώ Έχω ένα πρόβλημα με την ε, φράση «αναδυόμενες ε, προκλήσεις ασφαλείας». Θα ήθελα να, ε, να πω γιατί αναφέρομαι στο παρελθόν. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, η έσοδο επικεντρώταν σε επιθέσεις που αφορούσαν την τεχνολογία. Αυτό αναφέρεται στο βιβλίο, το βιβλίο του Κούκου, το αυγό του Κούκου ε, και ε, επιθέσεις που αφορούσαν χακαρίσματα. Αυτό ήταν, ήταν, ήταν ήδη από το 1986. όλο αυτό αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της γεωπολιτικής, γεωπολιτικής εδώ και πολλά χρόνια και αφορούσε τον ανταγωνισμό της εξουσίας. Η τεχνολογία αλλάζει, όμως οι σκοποί παραμένουν οι ίδιοι, οπότε η μεγάλη διαφορά είναι ο ρυθμός ε, με τον οποίο γίνονται αυτές οι αλλαγές και με τον οποίο οι απειλές εμφανίζονται και με βάση την αλλαγή την ταχύτητα των αλογών, η πραγματική πρόκληση ε, είναι η πολιτική ηγεσία, η διασυνδεσιμότητα μεταξύ των ε, συμβατικών μέσων διαμάχης και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Με άλλα λόγια, οι κυβερνοδράσεις ε, σχετίζονται με τις δράσεις των στρατευμάτων αλλά και με τις οικονομικές επενδύσεις και ο κοινό παρονομαστής είναι να εφαρμόσουμε μια γεωπολιτική στρατηγική. Με άλλα λόγια, έχει έρθει η ώρα να αλλάξουμε αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε το στρατηγικό ανταγωνισμό και τη διαμάχη στο μέλλον και να υιοθετήσουμε μια ολιστική προσέγγιση ε, στην ε, ανταπόκριση που θα έχουμε. Κυρίες και κύριοι, το 5G και η νέα τεχνολογία, σύρμα της τεχνολογίας θα ε, επιταχύνει την ε, τεχνητή νοημοσύνη, την ε, τεχνολογία, θα μεγαλώσει το εύρος ψηφιοποίησης της κοινωνίας, την, διεπαφή, την ανθρώπινη διεπαφή με τις επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα και τον πόλεμο και τις διαμάχες και σήμερα έχουμε μια ξεκάθαρη γραμμή μεταξύ της κυβερνοασφάλειας και της κυβερνοεπίθεσης. Όμως η, γραμμή αυτή δεν θα είναι τόσο ξεκάθαρη. Η εσωτερική ασφάλεια θα σταματήσει να εξίσει σε αυτό το πλαίσιο ή τουλάχιστον θα βασίζεται σε μερικές βασικές αξίες. Η ασφάλειά μας λοιπόν θα, θα βασίζεται κυρίως στην ψηφιακή υποδομή ε, και η ανταπόκριση των κυβερνήσεων και η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα θα είναι κάτι τόσο σημαντικό όπως και ο παραδοσιακός τομέας άμυνας η ανάπτυξη των δικτύων 5G αλλά και ε, η τεχνολογική εταιρεία Huawei ε, είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Προσφάτως ε, προτάθηκε ότι το δίκτυο 5G θα πρέπει να αναγνωριστεί ως στρατηγική επιλογή και όχι απλά τεχνολογική και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συντονίσει μια κοινή απάντηση ώστε να, να αντιμετωπίσει τους κινδύνους. Θα ήθελα να σας πω ότι η ιστορία έχει δείξει όταν, ότι όταν η Ευρώπη και η Αμερική συνεργάζονται είναι πιο ισχυροί. Όπως ε, ε, υπόθηκε πρόσφατα, το ΝΑΤΟ συνεχίζει να προσαρμόζεται για να μπορέσει να παραμείνει στο μέτωπο, να μείνει μπροστά στις νέες τεχνολογίες. Ε, συνεργαζόμαστε για να ενισχύσουμε την κυβερνοασφάλειά μας. Ο στόχος μας είναι να είμαστε τόσο αποτελεσματικοί στο κυβερνοχώρο, όσο είμαστε και στο έδαφος, στη θάλασσα και στον αέρα. Επικεντρωνόμαστε σε τεχνολογίες για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία. Από, από την άλλη πλευρά χρησιμοποιούμε τεχνολογίες της ε, στον τομέα της τεχνητή νοημοσύνης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε και να ε, επέμβουμε σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Επίσης, συνεργαζόμαστε με του συμμάχου μας. Ε, η κυβερνοασφάλεια αποτελεί κομμάτι της κοινή μα Άμυνα και μία επίθεση, κυβερνοεπίθεση επίσης μπορεί να ενεργοποιήσει το άρθρο 5. Επίσης δημιουργούμε δράσεις για την κυβερνοασφάλεια εδώ στη Μόνς, στο Βέλγιο όλα αυτά μπορούν να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, έχουμε χρησιμοποιήσει δυνατότητες ε, του κυβερνοχώρου κατά του ISIS ε, και αρκετές χώρες έχουν ε, προσφέρει τις κυβερνοδυνατότητες τους, μεταξύ των οποίων οι κάτω χώρες Αστονία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΙΠΑ. οι χώρες παραμένουν ιδιοκτήτριες αυτών των κυβερνοικονοτήτων όπως συμβαίνει και με τα οπλικά τους συστήματα θα ήθελα να ανασφερθώ σε αυτές τις επιτυχίες Πράγματι έχουμε δει ε, μια τρομερή συνεργασία ε, στην αντιμετώπιση απειλών, στην ανταπόκριση της ε, προσφυγικής κρίσης και συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία. Όμως το θέμα εδώ πέρα δεν είναι να προσθέσουμε και άλλα επίπεδα γραφειοκρατίας. Αντιθέτως, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται μια κοινή προσέγγιση και πόρους για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο και η συνεργασία ξεκινά με μια πολιτική συζήτηση όπως είναι αυτή οποία την οποία διεξάγουμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, αξιότιμη κύριε. Δεν έχουμε φτάσει στο τέλος, περιμένετε πριν χειροκροτήσετε. Έχουμε και έναν τρίτο εξαιρετικό μελετή και θα ακολουθήσει και συζήτηση. Κύριε Τόμας Βάλασεκ, από την Carnegie Europe. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω ενώπιον των μέλων του ε, Κοινοβουλίου. Αγαπητοί φίλοι, θα συνεχίσω ε, τα όσα είπα ο σας, όχι μόνο για να δείξουμε την ενότητα της Τσεχοσλοβακίας, αλλά διότι η τεχνολογία είναι ένα από τα πράγματα που εμείς υπεύθυνη λήψη αποφάσεων καταλαβαίνουμε λιγότερο. Συχνά αναρωτιόμαστε για τις διάφορε απειλέ ε, που έρχονται προς εμάς ε, υπό τη μορφή πληροφοριών, ε, ελλείψεων διαφόρων σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά σπάνια αναρωτιόμαστε πώς θα επηρεάσει τη δουλειά μας η τεχνολογική μεταβολή, οι τεχνολογικές αλλαγές. Το θέμα αυτό της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας ε, στον πόλεμο ε, είναι πολύ σημαντικότερο από τις παραδοσιακές απειλές. Ε, εστιάζομαι σε αυτό γιατί το καταλαβαίνει ο περισσότερος κόσμος λιγότερο. Πολλοί θα έχετε διαβάσει για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή θα επηρεάσει τον πόλεμο στο μέλλον, τη διεξαγωγή πολέμων στο μέλλον. Εγώ θα αλλάξω λίγο οπτική γωνία. Θα εστιάσω στην επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον της αμυντικής διπλωματίας. Ε, κάτι που απασχόλησε στη δουλειά μας και εμένα και τους συναδέλφους εδώ. Τι εννοώ όταν αναφέρομαι στην αμυντική διπλωματία υπό, αυτό το πρίσμα, πολύ απλό. Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγουν πολέμους ε, και επιχειρήσεις οι ευρωπαϊκές χώρες είναι ομαδικός συνήθως. Ε, σπάνια χώρες του ΝΑΤΟ ή της Ευρώπης διεξάγουν πόλεμο μόνες τους. Ωστόσο, η διεξαγωγή πολέμου ε, με συντονισμένο τρόπο δεν είναι κάτι παρα... κλασικό. Κάθε κράτος έχει άλλη ιστορία, ε, χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του διαφορετικά, ε, κλασικά, παραδοσιακά και βλέπει τι επιχειρήσεις διαφορετικά. Ο λόγος για τον οποίο διεξάγουμε μαζί διάφορες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ως ΝΑΤΟ είναι ότι έχουμε θεσπίσει διάφορες διαδικασίες κανόνες, ε, βήματα πολύ συγκεκριμένα, ώστε να διατηρούμε την ενότητά μας. Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούμε από κοινού ε, πληροφορίες, τις οποίες αξιολογούμε με τον ίδιο τρόπο. Όχι όλοι, αλλά προσπαθούμε με κάποιο τρόπο αντιπροσωπευτικό να τις ερμηνεύουμε, σαν να ήταν η ερμηνεία και των 28 χωρών. Ε, ασκούμε πολιτική επίβλεψη, υποπτία όλων των επιχειρήσεων δεν εμπιστευόμαστε απόλυτα τους στρατιωτικούς διοικητές, αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι και οι 28 χώρες έχουν να πούν κάτι, λαμβάνοντας υπόψη τις ε, τοπικές ευαισθησίες κάθε χώρας ε, για κάθε επιχείρηση. Οπότε για κάθε επιχείρηση η πίεση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τον e ΕΚ στο πλαίσιο της Ατλαντικής ε, Συμμαχίας έχουν να πούν κάτι. φροντίζουμε να συμφωνούμε για τις απαιτήσει όσον αφορά τον εξοπλισμό μαζί εκ των προτέρων, ε, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ανησυχίες των μικρότερων κρατών. Μελών επίσης. Θα μπορούσα να συνεχίσω επάπειρον, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι φυσικό 28 ή 29 χώρες όπως το ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διεξάγουν επιχειρήσεις μαζί. Ο λόγος για τον οποίο τα καταφέρνουμε και ο λόγος για τον οποίο η εχθροί μα δεν έχουν καταφέρει να μας ε, διαιρέσουν, δεν είναι ότι δεν προσπάθησαν, είναι ότι εμείς ε, στη διεξαγωγή των επιχειρήσεων έχουμε αυτή τη συνένεση, ε, την οικοδόμηση εμπιστοσύνη και τη σχετική διαδικασία. Πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη όλα αυτά και για ποια είναι η τεχνολογική πτυχή του ζητήματο απλό. διάφορε τεχνολογικέ απειλέ υπάρχει ε, κίνδυνος να ε, καταλύσουν ε, όλα αυτά που έχουμε χτίσει την τελευταία 20 αιτία. Πώς και τι. Οι βασικές τάσεις που με απασχολούν είναι η εμφάνιση του αυτοματοποιημένου πολέμου. Το ότι μπορεί ο πόλεμος στο μέλλον να διεξάγεται από drones που θα λειτουργούν από απόσταση, με έλεγχο από απόσταση, αλλά και έξυπνα θα μαθαίνουν δηλαδή από τα δικά τους λάθη και αυτόματα θα προσαρμόζουν τις τακτικές τους ε, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Δεν επικρίνω εδώ τώρα την ορθότητα του ζητήματος κατά πόσο είναι σωστό ή λάθος, αλλά ξέρω από τη δική μου έρευνα ότι πολλές ε, ε, χώρες της Ευρώπης έχουν προχωρήσει πολύ στην έρευνα αυτής της τεχνολογίας. Δεν παρακολουθούμε απλά τα όσα γίνονται στην Κίνα και στις ΗΠΑ. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες ήδη έχουν αναπτύξει ή αναπτύσσουν την τεχνολογία αυτή. Και το λέω τώρα αυτό διότι ενδέχεται να υπάρξει παγκόσμια απαγόρευση στο εγγύς Και πάλι εδώ δεν είναι εκτίμηση αυτό που λέω. Ο αυτοματοποιημένος πόλεμος, το θέμα δεν είναι εδώ αν είναι σωστός ή λάθος, είναι ότι δεν υπάρχει απόλυτη συνένεση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, οπότε Ωστόσο, μπορεί η τεχνολογία να εμφανιστεί πριν ληφθεί η απόφαση απαγόρευσή τη. Αυτή η τεχνολογική τάση στην οποία αναφέρομαι, πώς θα εξελιχθεί η, η πιθανότητα σμήνει ε, drones να διεξαγούν τους πολέμους στο μέλλον και πώς αυτό επηρεάζει του, όλους εμάς ουσιαστικά βγάζουν τον άνθρωπο από την εικόνα και επιταχύνουν τρομακτικά τις ε, επιχειρήσεις. Ε, επιχειρήσεις που θα χρειάζονταν ώρες, ημέρες, εβδομάδες, ε, αν χρησιμοποιούσαν ανθρώπους, θα χρειάζονται λεπτά, ώρες το πολύ. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο δεν θα έχουμε ξαναδεί και θα επηρεάζει τα πράγματα με τρόπους που δεν θα ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε ε, ως θεσμοί. Πρώτον, πώς μπορούμε να ασκούμε πολιτική εποπτεία σε επιχειρήσεις όταν οι επιχειρήσεις ε, διαρκούν λεπτά ή ώρες. Δεν έχουμε τέτοια συνηθίσει κάτι τέτοιο. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ συνήθως χρειαζόμαστε έγκριση των διοικητών μας ε, λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουμε μια επιχείρηση και μετά πριν κάνουμε οτιδήποτε σημαντικό ζητάμε την έγκρισή τους πάλι. Αυτό δεν θα είναι εφικτό σε επιχειρήσεις που διαρκούν λεπτά ή ώρες. Η εμπιστοσύνη λοιπόν των κρατών και των πολιτών σε αυτή την τεχνολογία θα υπονομευτεί. Τώρα για τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη η ενότητα μεταξύ των κρατών μελών επίσης θα είναι πιο δύσκολη. Διότι μόνο λίγες χώρες αναπτύσσουν αυτή την τεχνολογία, είναι εξαιρετικά περίπλοκη, εξαιρετικά ακριβή, απαιτεί τη δυνατότητα να συγχωνεύει κανείς ε, με αρκετά προχωρημένο τρόπο πολλέ ε, ε, προηγμένες τεχνολογίες, αλγόριθμους, λογισμικά και μόνο λίγες χώρες θα τα καταφέρουν. Αντίθετα από το ΝΑΤΟ, δεν έχουμε τον ίδιο διαμερισμό ε, βαρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τη είπα. Δεν αφιερώνουμε πάνω από το 2% στις αμυντικέ δαπάνες, όπως είπα αλλά και λίγε χώρε ε, έχουν την τεχνολογία που απαιτείται. Οι υπόλοιπε χώρε δεν την διαθέτουν. Οπότε αντιλαμβάνεστε πώ αυτό θα δυσκεράνει ε, τι ενδοευρωπαϊκέ μα σχέσει. Τρίτο, τι γίνεται όσον αφορά την εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών σε περίπτωση που η τεχνολογία δεν συμπεριφέρεται όπως θέλουμε. Ε, και στην εκμάθηση μηχανημάτων και στην τεχνητή νοημοσύνη υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα μηχανήματα θα προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους ε, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ε, μαθαίνοντας από τα δικά τους λάθη. Κανένα διοικητή δεν θα υπάρχει ο οποίο θα μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τι ακριβώς θα κάνει η τεχνολογία, τι ακριβώς θα κάνει το μηχάνημα κατά τη διάρκεια μιας επιχείρηση. Πώς λοιπόν να δείξουμε εμπιστοσύνη σε έναν διοικητή και πώ να αναθέσουμε ε, την ευθύνη σε ένα διοικητή να διεξάγει μια τέτοια επιχείρηση αν ο ίδιος δεν είναι πλήρω ε, ικανός να μας εξηγήσει τι θα γίνει κατά τη διάρκεια τη επιχείρηση. Ε, και υπάρχουν και άλλα πολλά επιχειρήματα. Το θέμα είναι ότι όσο αλλάζει η φύση του πολέμου και όσο περισσότερο βασιζόμαστε σε μηχανήματα και όσο και περισσότερο οι εχθροπραξίε διαρκούν λεπτά και όσο περισσότερο η τεχνολογία είναι το κλειδί του πολέμου στο μέλλον, και όσο λιγότερα τα κράτη-μέλη που θα διαθέτουν την τεχνολογία, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να ακολουθούμε τι διαδικασίε που είχαμε στο παλιά, να λαμβάνουμε αποφάσει ω 27, 28, 29 κράτη-μέλη. Και δεν θα έχουμε το χρόνο να αποφασίζουμε και να εγκρίνουμε κάθε στάδιο τη επιχείρηση. Ε, κάτι θετικό. Καμία από τις δυσκολίες ε, που ανέφερα δεν είναι ανυπέρβλητες. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου ε, τα τεχνολογικά θέματα ή τα διπλωματικά μπορούν να επιληθούν. Ε, για παράδειγμα, μπορεί να οικοδομηθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ε, σε συνεργασία μεταξύ μη στρατιωτικών και στρατιωτικών δυνάμεων ώστε όλοι να καταλαβαίνουν απόλυτα τι κάνουν τα μηχανήματα. Ένας τρόπος ε, είναι οι ασκήσεις, οι δοκιμές. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε προσωμιώσεις εχθροπραξιών και εκπρόσωποι κρατών μελών να ζητούν προσωμιώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση ή ΝΑΤΟ πριν δώσουν την άδεια σε στρατιωτικούς διοικητέ να διεξάγουν κάποιε επιχειρήσει. Ένα άλλο μέτρο το οποίο θεωρώ σημαντικό και πιστεύω θα γίνει σύντομα θα ήταν ένας έλεγχος των σημερινών μας προτεραιοτήτων σε θέματα εξοπλισμών ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι μπορούν να εγκριθούν. Να σα θυμίσω μια εμπειρία ενός πρόσφατου πολέμου που στις αρχές του πολέμου ε, τα τεράστια ε, καταδρομικά με πολύ μεγάλα όπλα πάνω τους θεωρούνταν η καλύτερη τεχνολογία και πολύ ε, σύντομα θεωρήθηκαν απερχαιωμένα και τα αεροπλανοφόρα πολύ γρήγορα πήραν τη θέση τους και κυριάρχησαν ε, τις επόμενες δεκαετίες. Το ίδιο μπορεί να συμβεί τέτοια γρήγορη αλλαγή με κάποιες ε, πλατφόρμες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες ε, όπως είναι τα αυτόνομα drone. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα μεταβάλουν τις ε, μελλοντικές μας ικανότητες και τις προτεραιότητές μας. Τέλος, όλο αυτό το πρόβλημα είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Πολύ δύσκολο για τους περισσότερους από μας ε, όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. Ε, δύσκολο να το καταλάβουμε. Ε, το λεξιλόγιο, οι γνώσεις ε, μας λείπουν για να καταλάβουμε επαρκώς τις τεχνολογικές προκλήσεις. Ελάχιστοι από εμά γνωρίζουμε τα τεχνολογικά θέματα, οπότε το καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ για όσον αφορά αυτή τη μελλοντική τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο είναι να γίνονται περισσότερε ενημερώσει, περισσότερη πληροφόρηση, περισσότερε συζητήσει. Να εξετάζουμε τι δυνατότητε όχι μόνο για το μέλλον ε, του πολέμου, αλλά και για το πώ θα επηρεάσει αυτή η νέα γενιά πολέμου εμάς. Ε, θα πρέπει από τώρα να εξοικειωθούμε με το λεξιλόγιο, με τις πιθανές προκλήσεις, να, ώστε να μην βρεθούμε σε μειονεκτική θέση, διότι οι λαοί μας και η ελίτ μας δεν γνωρίζουν τι ακριβώς θα συναντήσουμε και αν ε, επιλέξουμε μια τέτοια οδό θα είναι δύσκολο να διασφαλίζουμε συμφωνία 28-29 κρατών στον τομέα αυτών των τεχνολογιών ε, όταν κάποια κράτη-μέλη θα έχουν λιγότερες ηθικές ε, επιφυλάξεις από άλλα και θα μας θέσουν σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα, ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση. Αυτά και είμαι έτοιμος να απαντήσω ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Αρχίζει τώρα η συζήτηση. Η Κλέρ Μούντι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Και το τελευταίο για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι τεχνολογίες πραγματικά εξέλισσονται ραγδαία και θα πρέπει να δούμε πώς θα ρυθμίσουμε τη συνέχεια για νομοθετικά. Έχω πολλές ερωτήσεις προς πολλές κατευθύνσεις, ακριβώς γιατί είναι και τόσες πολλές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Και έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για μια νέα φάση των παγκοσμίων ε, σχέσεων. Γιατί ιστορικά έχουμε εστιαστεί στις βασικές προκλήσεις και αυτές οι προκλήσεις τώρα όλο και περισσότερο έρχονται κατά πάνω μας από διάφορες κατευθύνσεις και γωνίες και εσωτερικές είναι. Ε, συμφωνώ για τη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και πόσο σημαντικό είναι αυτό. Ε, ε, θα πρέπει να τα βλέπουμε σφαιρικά τα πράγματα. Και δεν μιλήσατε όχι μόνο για την πρακτική προσέγγιση, αλλά και για την πολιτική, διότι επιπτώσεις ορισμένων τουλάχιστον από τις απειλές αυτές αφορούν και τις δικές μας πολιτικές και τις επηρεάζουν. Το έχουμε δει αυτό και θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε μέχρι να ε, αποκτήσουμε ε, συντονισμένη και αποτελεσματική απόκριση στις απειλές αυτές και στις πολιτικές ε, παρεμβάσεις που βλέπουμε για τη Μέση Ανατολή. Ε, έχουμε τη Μέση Ανατολή, το Ανατολικό Μέτωπο, το κυβερνοπόλεμο, τις νέες τεχνολογίες και ποιος ξέρει ποιες θα είναι αυτές και τι θα αντικαταστήσουν. Και είναι μπροστά μας πραγματικά και οι γεωπολιτικές δομές κτλ. Κάτι που δεν ανέφερε κανένα σας όμως είναι η πυρηνική απειλή. Που νομίζω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να την παραμελήσουμε. Τώρα βλέπουμε τη συμφωνία για τα όπλα αμέσου ελληνικούς, ε, όπου και τα κράτη-μέλη της Ευρώπης έχουν ε, συνυπογράψει, αλλά εμείς είμαστε οι κύριοι δικαιούχοι. Και τώρα απειλείται αυτή η συμφωνία. Ε, και οποιαδήποτε απειλή αυτή θα μπορούσε να είναι ολέθρια δεν θέλουμε να ξαναδούμε τα πυρηνικά να γίνονται τόσο περίπλοκο θέμα, γιατί είναι και πολύ περισσότερες οι χώρε από τότε που υπεγράφει η συμφωνία για του πυράβλου μέσου ελληνικού. Άρα, ε, περιμένω πραγματικά τις απαντήσεις σας, να δούμε πώς μπορούμε στο μέλλον να ρυθμίσουμε τα θέματα των πυρηνικών όπλων για να αντιμετωπίζουμε και την πυρηνική απειλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Θα πρέπει όμως να γίνει μια διάκριση μεταξύ των πολιτικών ομάδων. να <laughs> μην δώσω το λόγο σε δύο, δηλαδή ταυτόχρονα από την ίδια πολιτική ομάδα. Ο κύριος Κούκαν θέλει το λόγο. Όχι. Ε, τότε ο κύριος Πάσκου. Απουσία των μαχητών, ο πόλεμος αναβάλλεται, έτσι, μάλλον γι' αυτό παίρνω εγώ το λόγο μετά την Κλέρ Μούντι. Νομίζω ότι θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε αυτά που είπε ο κύριος Βάλασεκ. Διότι μέχρι τώρα ο, κο... ο πόλεμος ήταν ένα θέμα που είχε πάρα πολύ μεγάλη ένταση εργασίας. Αν δείτε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ε, βλέπετε πόσες ένοπλες δυνάμεις είχαν εμπλακεί και πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και το ένα και το άλλο. Τώρα όμως, ποιο είναι το παράδοξο. Οι χώρες εκείνες οι οποίες έχουν πάρα πολλές δυνάμεις, θέλουν, ένοπλες, θέλουν να τις αντικαταστήσουν από μηχανές. Και οι άλλοι που δούλευαν σε ένοπλες δυνάμεις, τι θα γίνουν, άνεργοι. Δεύτερη ερώτηση. Ο πόλεμος αναπόφευκτα έχει μια αρνητική επίπτωση ε, και εξισορρόπησης των πληθυσμών. Τώρα τι θα γίνει αν δεν σκοτώνεται κανένας, αν σκοτώνονται μεταξύ τους τα ρομπότ. You asked, Mr. very... Κύριε Βαλασέκ, έθεσατε μια πολύ εύστοχη ερώτηση. Πώς θα παίρνεις αποφάσεις και ποιος θα αποφασίζει και τι θα αποφασίζει. Πώς θα ε, αναπτυχθούν δεν ξέρω τι σμήνει drones ή άλλων οπλικών συστημάτων. Αυτές θα είναι οι αποφάσεις. Τα πάντα αλλάζουν. Και όσο νωρίτερα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τις επιπτώσεις όλων αυτών, τόσο το καλύτερο. Πρώτα με τα think tanks, τις ε, εξαμενές σκέψεις και τις ομίλους προβληματισμού και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέσβη, κύριε Σεράνο, ξέρετε ότι ελπίζω να μην αναθέσουμε και τη διπλωματία σε μηχανές, ότι να τεκλιτώσει οι διπλωμάτες να παραμένουν σημαντικοί στο μέλλον. Αλλά καθόλου βέβαιο και αυτό. Εγώ δεν ξέρω τι είδου αλγόριθμοι ε, θα μπορούσαν να συμμετέχουν για να κάνουν στην άκρη και τη διπλωματία. Και τελειώνω με αυτό. Πραγματικά έχει έρθει η ώρα να καθίσουμε και να προβληματιστούμε πάρα πολύ σοβαρά για όλες αυτές τις εξελίξεις. Ευχαριστώ. Thank you. Um... Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ακολουθήσω την ε, παρουσίαση του κύριου Πασκού. και θα ήθελα να ρωτήσω όλους τους ε, συμμετέχοντες, όλους τους προσκεκλημένους ήταν ένας ε, γνωστός τομέας ε, το ότι γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι ακόμα έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε πάνω σε αυτό το τομέα ε, και γι' αυτό το λόγο μου έκανε εντύπωση η παρουσίαση του προσβευτή Σεράνο. Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω όλους τους ομιλητές ποιες δράσεις ε, πρέπει να ληφθούν τους ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές. Ίσως να ακούγεται φιλίς αυτή η ερώτηση, όμως όπως και να έχει πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε να το σκεφτόμαστε Αυτός ήταν, αυτό ήταν το τέλος των ερωτήσεων και θα ακολουθήσουμε την ίδια σειρά με προηγουμένους. Ο κύριος Σεράνο, ευχαριστώ πολύ που ε, αναφέρατε ε, το ζήτημα των πυρηνικών αλλά και της τεχνητής ε, νοημοσύνης που είναι πολύ σημαντικά θέματα. Πριν όμως απαντήσω πάνω σε αυτό θα ήθελα να θέσω το ρητορικό ερώτημα σε ε, τι βαθμό τα ερωτήματα αυτά θα επηρεάσουν τις διαμάχες που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα στην περιοχή του Σαχέλ, όπου αύριο συγκεκριμένα θα μεταβώ στο Τσάντ. Θα έλεγα ότι το, τα πυρηνικά ζητήματα δεν έχουν κανένα ρόλο εδώ πέρα. Η τεχνητή νοημοσύνη τώρα έχουμε δει ότι σε πολλές από αυτές τις ε, διαμάχες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα στην Αφρικανική Ήπειρο η υψηλή τεχνολογία δεν έχει φτάσει εκεί ακόμα. Ναι, ίσως ε, ναι, θα γίνει πιο ε, φθηνή, θα επεκταθεί περαιτέρω, όμως πιστεύω ότι ακόμα για, μεγάλο, για μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα. Και ένα σχόλιο το οποίο ήθελα να τονίσω είναι ότι ε, ε, στην πραγματικότητα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές ε, διαμάχες, όμως δεν αφορά την μάχη αυτή καθ' αυτή, αλλά αφορά περισσότερο την διαδικασία της συμφιλίωσης. Και πιστεύω ότι ως διπλωμάτες αυτός είναι ο ρόλος που θα πρέπει να εκπληρώσουμε. Με βάση ε, την ανάλυση ε, του ποιες είναι οι πηγές έντασης ε, και διαμάχης. Ναι, οι μηχανές, η τεχνολογία είναι πολύ σημαντικά θέματα. Όμως εν τέλει το κλειδί επίλυσης της διαμάχης είναι τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε. Ποιοι είναι οι στόχοι μας και για ποιο λόγο ξεκινά μία διαμάχη. Για ποιο λόγο υπάρχει ο ανταγωνισμός θα ήταν εύκολο να πούμε, ε, να εξηγήσουμε ότι μπορεί να υπάρχουν περιφερειακές ε, διαμάχες σε κάποιες περιπτώσεις ε, ή κρατικές δομές που δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικά τον πληθυσμό που κυβερνούν. Αυτά είναι κάποια προβλήματα. Μετά έχουμε ένα άλλο πρόβλημα που αφορά τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Και εδώ πέρα λοιπόν εισερχόμαστε σε ένα διαφορετικό ε, πλαίσιο, σε διαφορετικό παιχνίδι διότι εν τέλει αυτός ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, παρόλο που υπάρχουν και άλλα ε, στοιχεία, όχι μόνο αυτό το θέμα της άμυνας, αλλά και το βιομηχανικό, το οικονομικό και αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία και συνδέονται μεταξύ τους σε ένα βαθμό με την ανάπτυξη των όπλων έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικές κατηγορίες διαμαχών και πιστεύω ότι ο μεγάλος ανταγωνισμός ε, θα σχετίζεται περισσότερο. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν και τα άλλα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όπως και να έχει λοιπόν το σημαντικό είναι να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε, ποια πρόκληση υπάρχει. Η διπλωματία λοιπόν δεν νομίζω ότι θα ανταγωνιστεί από ε, μηχανήματα. Όταν το είπατε αυτό, σκέφτηκα το Star Trek. Έχουμε μηχανήματα για τον πόλεμο. Όμως το ενδιαφέρον είναι ότι στο Star Trek πάντοτε υπάρχουν διπλωμάτες ε, που είναι άνθρωποι ή όντα που έχουν ανθρωπόμορφα όντα που πάντοτε προσπαθούν να βρουν μια λύση ε, στις ε, διάφορες ερμηνείες της εκάστοτε πραγματικότητας και προσπαθούν να βρουν λύσεις. Ε, καθότι και εγώ είμαι διπλωμάτης, ελπίζω ότι δεν θα αντικατασταθώ από μηχανήματα. Όσον αφορά το πυρηνικό κομμάτι, το έχουμε την τάση να το ξεχνάμε, όμως το INF ήταν ένα πολύ ισχυρό ε, μήνυμα και θα ήθελα να σας πω ότι ε, η ε, αποπυρηνικοποίηση θεωρεί, συνεχίζει να είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Η πυρηνική αποτροπή επίσης παίζει έναν σημαντικό ρόλο παγκοσμίως, όμως θεωρώ ότι υπάρχει ε, μια, ένα σημαντικό θεματολόγιο πάνω σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ιδιαίτερο την ε, μη διάδοση και τον αφοπλισμό. Του χρόνου ε, θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και πάλι. το οποίο θα αποτελέσει ένα σημαντικό στοιχείο της διεθνούς μας ατζέντα και θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το ε, ζήτημα των ε, πυρηνικών ε, βελληνικού. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το πώς αυτό θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και να αντιμετωπίσουμε με μια πιο παγκόσμια προσέγγιση και ναι υπάρχουν ε, σκέψεις πάνω σε αυτό και στην ΕΙΕΔ. Δεν έχουμε ξεχάσει λοιπόν αυτό το σημαντικό στοιχείο, όπως επίσης δεν ξεχάσαμε και την τεχνική, τεχνητή νοημοσύνη που επίσης είναι πολύ ψηλά στο θεματολόγιο μας και θα ε, εξετάσουμε αυτά τα θέματα. Θα εξετάσουμε τις, ε, τους κανόνες πάνω στους οποίους πρέπει να προσαρμόζονται όλα τα όπλα την ε, συλλογή των κανόνων που ρυθμίζουν ε, τον, ε, το ζήτημα των, των πολεμικών σειράξεων, το ζήτημα της αναλογικότητας και θα δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Το σημαντικότερο θέμα βέβαια σε όλες αυτές τις συζητήσεις, όπως γνωρίζετε, είναι ο ανθρώπινος παράγοντος να παραμένει ε, στην ε, λήψη των ε, αποφάσεων. Φυσικά όσοι εξετάζουν αυτά τα συστήματα θα θέλουν να διασφαλίσουν ότι η σκανδάλη βρίσκεται σε ανθρώπινα χέρια Οι άνθρωποι βέβαια ποτέ δεν ήταν ε, ένας, ε, ε, μία εγγύηση, όμως σίγουρα καλύτερα να είναι ένας άνθρωπος παρά μία άβουλη μηχανή που έχει κατασκευαστεί από άνθρωπο. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε εγγυήσει και μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν λοιπόν ότι δεν θα δημιουργηθεί ένα τέρας το οποίο δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε. Και φυσικά υπάρχουν σκέψεις και συζητήσεις πάνω σε όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν που παρουσιάσατε αυτές τις σκέψεις. Ευχαριστώ πολύ για το έργο σας τα τελευταία πέντε χρόνια και θα χαρώ πολύ να συνεργαστώ μελλοντικά με πολλούς από εσάς και ευχαριστώ επίσης ε, όλους όσους ε, ε, με βοήθησαν και συνεργαστήκαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη και Χαβράνεκ. Ευχαριστώ για τα πυρηνικά όπλα. Ευχαριστώ που το θίξατε. Ναι, υπάρχουν πράγματι. Και η σχετική άμυνα εναντίον πυρηνικών όπλων είναι σημαντικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Τώρα για τη συνθήκη INF για τα πυρηνικά μεσοβελληνικούς μετά από το ψυχρό πόλεμο υπήρχαν περίπου 3.000 ε, ε, πύραυλοι πυρηνικοί μεσοβελληνικούς και απαγορεύτηκαν από όλους, από τη συνθήκη αυτή, όλοι αυτοί. Ήταν πολύ αποτελεσματικό, αλλά η Ρωσία παραβίασε τη συνθήκη με το συστημα ssc SSE8, ε, το οποίο επίσης είναι πυρηνικό και ως αποτέλεσμα οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να αποσυρθούν από τη συνθήκη αυτή. Έχει ακόμα περιθώριο να συμμορφωθεί η Ρωσία, αλλά καλό θα ήταν να ετοιμαζόμαστε για έναν κόσμο χωρίς τη συνθήκη ΑΕΝΕΦ. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανταπαντήσουμε, να ξεκινήσουμε έναν ε, εξοπλιστικό αγώνα ή κάτι τέτοιο. Αλλά όπως είπε ο κύριος Σεράνο, πρέπει να δούμε καθολικά και σε παγκόσμιο επίπεδο το ζήτημα αυτό. Ο περιορισμός των ε, όπλων, ο έλεγχος των όπλων από τον ΝΑΤΟ είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει ήδη να ξεκινήσουμε έναν διάλογο με τη Ρωσία για το θέμα αυτό. Και έχουμε κοινοποιήσει τις προθέσεις του ΝΑΤΟ πολύ σαφώς. Η μη τήρηση αυτή τη συνθήκη όμω από την πλευρά τη Ρωσία είναι σημαντικό πλήγμα για το σύστημα αυτό ελεγχού όπλων. Οπότε πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με τρόπο αποτελεσματικό. Τώρα το πιο φιλοσοφικό ερώτημα της σχέσης μεταξύ της ανθρωπότητας και των μηχανημάτων. Την απάντηση μπορεί κανείς να βρει στην ιστορία, στις αιτίες κοινωνικών αταραχών στο παρελθόν, να δούμε τα πράγματα που προκάλεσαν μεγάλη αποσταθεροποίηση αν όχι και στη λογοτεχνία το 1920 ο Κάρο Τσάπεκ ε, τσέχος ε, ε, συγγραφέας και θεατρικός συγγραφέας έγραψε ένα θεατρικό έργο που περιγράφει μια ιστορία ρομπότ που καταλαμβάνουν τον κόσμο αφού δημιουργήθηκαν από τους ανθρώπους είναι σαν μια ειδοποίηση 100 χρόνια αργότερα θα μπορούσε να αποτελεί πηγή έμπνευση για να βρούμε απαντήσεις στα ερωτήματα που κάνατε εσείς εδώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν και ξανά, ξανά και ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βάλασεκ. Ευχαριστώ και πάλι που ε, ε, μου δίνετε το λόγο εξαιρετικά τα ερωτήματα για το θέμα της πυρηνικής απειλής συμφωνώ απολύτως ε, με τα όσα είπε ο πρέσβης Σεράνο ότι κυρίως εδώ ασχολούμαστε με συμβατικά όπλα, αλλά έχουμε φυσικά και συμφέρον ως κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ζούμε σε ένα κόσμο που θα επιδίδεται σε μια κούρσα εξοπλισμών ε, και αυτό κοστίζει και πόρους κτλ. Η στρατηγική ε, ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει προθυμία ε, γιατί υπάρχει και μεγάλη δυσπιστία μεταξύ των κρατών μελών. Ε, τα πράγματα μάλλον θα χειροτερέψουν πάρα πολύ πριν βελτιωθούν. Δεν βλέπω πολιτική βούληση αυτή τη στιγμή για διαπραγματεύσεις ε, ουσιαστικές. Τώρα μπαίνουμε σε μια νέα συζήτηση για τη στρατηγική σταθερότητα και έχει κάνει και η δουλειά το Κάναγκη. Θα πρέπει να είναι πολύ διαφορετική συζήτηση από τις συζητήσει για τις συνθήκες του 70 για τη μη διάδοση των πυρηνικών και για τους πυράβλους μεσοβελληνικούς. Ε, έχουμε πυράβλους τώρα συμβατικούς με μεγάλη ακρίβεια και μπορούν να κάνουν και μεγάλη ζημιά και με μεγάλη, ε, μεγάλη ευνηδιαστική ε, δράση. υπάρχουν ε, υπερηχητικοί υπερακριβείς πύραυλοι των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν είναι τελείως τρελή η Ρωσία που ανησυχεί. Η μία πλευρά μπορεί να παραλύσει ε, τις ε, πυρηνικές κεφαλές της άλλης με ε, κυβερνοεπίθεση και θα πρέπει να είναι ε, τμήμα της ε, εξίσωσης και αυτό το στοιχείο να αναγνωρίσουν και να υπογράψουν και δύο πλευρές ότι δεν θα επιτεθούν στον κυβέρνο κέντρο διοίκησης των, των πυράβλων. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, λέγουν ότι σταμάτησε η Ρωσία να τηρεί τη συμφωνία ΕΝΕΦ λόγω της Ρωσίας και του οπλοστασίου. Οι Ρώσοι θα σας πούν το αντίθετο. Ότι θέλουν το ελεύθερο για να αναπτύξουν πυράβλους μεσοδελληνικούς κατά της Κίνας. Ε, δεν λέω ε, τι έχει κάνει η Κίνα, δεν ξέρω αν έκανε τίποτα κακό. Αλλά οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, αποσύρονται γιατί δεν τηρεί τη συμφωνία η Ρωσία. Πάντω και οι δύο πλευρές ανησυχούν πολύ μάλλον για την Κίνα αυτή τη στιγμή και δεν ε, μπορεί να υπάρξει ε, στρατική συμφωνία που να παραγνωρίζει την Κίνα. Έχω ζήσει μια εβδομάδα, ήμουν στο Πεκίνο και στο μέλλον δεν φαντάζομαι να αλλάξει τη βασική φιλοσοφία ότι <laughs> είμαστε μικρή αναπτυσσόμενη χώρα, αυτά είναι ζητήματα που αφορούν τις μεγάλες ανεπτυγμένες χώρες και μην μας ενοχλείτε με αυτή. Ε, και πάλι για τις μηχανές και τα ρομπότ και τον πόλεμο. Συμφωνώ με τον πρέσβη Σεράνο. Θα, δεν θα χαθούν οι διπλωμάτες, όχι απλώς επειδή ήμουν μέχρι πρόσφατα και εγώ διπλωμάτης, αλλά η ιδέα ότι μπορούμε να ελέγξουμε ε, την κατάσταση και να έχουμε παντού ανθρώπινη παρουσία πρέπει να ε, επανεξεταστεί. Γιατί εκείνοι που θα επιλέξουν να βγάλουν τον άνθρωπο και να ποντάρουν 100% στη μηχανή θα έχουν τεράστιο ε, πολεμικό και στρατηγικό και αμυντικό πλεονέκτημα που θα χάσουμε εμείς εάν διατηρούμε τον άνθρωπο. Αυτό ακούγεται έτσι κάπως φοβιστικό, μας τρομάζει. Αλλά ε, αν πάμε στη μικροδιαχείριση ε, της στρατιωτικής επέμβασης είναι ένα τελείως νέο φαινόμενο. Παλιά στέλναμε κανονιοφόρους, με ε, διάφορα εφόδια να, να πολεμούν τον κόσμο και δεν επικοινωνούσαν ε, και ελπίζαμε να τους ξαναδούμε και συχνότερα, μάλλον τις περισσότερες φορές δεν τους ξαναβλέπαμε. Ε, υπερβάλλω, αλλά θα πρέπει ως άνθρωποι και διπλωμάτες του μέλλοντος να συμφιλειωθούμε με την ιδέα ότι θα δώσουμε λίγο ε, από τον έλεγχο στις μηχανές. Δεν ε, θα πρέπει έτσι με αιμονή να θέλουμε να ελέγχουμε κάθε στάδιο ε, της μικροδιαχείρισης. Μπορεί αυτό να είναι ενοχλητικό και δύσκολο να το δεχτεί κανείς, είναι πραγματικότερο. Προσπάθησα στην εισαγωγή να σας πω τι πρέπει να κάνουμε, όπως ζήτησε η Πρόεδρος. Ε, θα πρέπει να ελέγξουμε και λογιστικά τις ε, δυνατότητές μας, τις ικανότητές μας και να μην σπαταλάμε δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς που μετά από 10 χρόνια θα είναι απαρχιωμένοι. Και εκπαίδευση για την τεχνητή νοημοσύνη. Ασχολείται ήδη, Πατή εκπρόσωπος, είναι καινούρια. Υπάρχουν και θέματα δεοντολογίας της τεχνητής νοημοσύνης ασχολείται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτά. Δεν ξεκινάμε από μηδενική βάση, αλλά θα πρέπει να διευρυνθεί ε, η κοινότητα ε, εκείνων που ασχολούνται με αυτά τα θέματα της ε, τεχνητής νοημοσύνης. Να προσθέσω και δύο-τρία άλλα σχόλια, μια που τελειώνουμε εδώ. Η σύμμαχοι που αναπτύσσουν αυτή την τεχνολογία θα πρέπει να ενημερώνουν τα άλλα κράτη-μέλη που δεν την έχουν για την ηθική, τη διεντολογία και πώς δουλεύει. Για τον εξής απλό, απλό λόγο. Αν είμαστε σε μια κατά, ε, ε, κατάσταση που χρησιμοποιούμε ε, τεχνητή νοημοσύνη, οι αντίπαλοι μας θα χρησιμοποιήσουν τη δική μας άγνοια για να μας φέρουν αντιμέτωπους ε, τα κράτη που έχουν την τεχνολογία και την καταλαβαίνουν απέναντι σε ε, ε, κράτη που δεν έχουν την τεχνολογία και δεν την καταλαβαίνουν. Τα περίφημα ρομπότ δολοφόνοι, αυτά τα killer robots δηλαδή, θα πρέπει να είναι σε γνώση όλων μας. Εγώ δεν ζητάω τον κώδικα, ούτε την, τις τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά τι σημαίνει για μας τι σημαίνει για τους άλλους και πώς γίνεται αυτό με την αμυντική διπλωματία για να μην μας διχάζουν οι αντίπαλοι μας. Θα μπορούσαμε επίσης να έχουμε και περισσότερη ενότητα για την ηθική και τη διοντολογία. Είναι πολύ σημαντικό ε, όσο ε, είμαστε διηρεμένοι εκεί για τον αυτόνομο πόλεμο, γιατί και πάλι οι αντίπαλοι μας θα προσπαθήσουν να, διχάσουν τα κράτη-μέλη. Ε, ξέρουν ότι χρειάζεται και ομοφωνία. Υπενήχθηκε ο Πρέσβη Σεράνο ότι γίνεται δουλειά. Υπάρχουν επιχειρήματα κατέρωθεν υπέρ και κατά ε, της αυτόνομης εξαγωγή των μαθών. Όταν έχει ένα 18χρονο ενθουσιασμένο με ένα joystick και, ε, που πίνει καφέδες όλη μέρα καφέινη, ε, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ο καταλληλότερος για να πάρει την απόφαση επειδή είναι άνθρωπος. Ε, έχουμε εκπάθηση από μηχανές, ε, περιορισμένη προς το παρόν, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια πολύ καλή ισορροπία. Πάντως χρειάζεται οπωσδήποτε συμφωνία σε επίπεδο 27 ή 28 για τη διαδολογία της τεχνολογίας και της χρηστής. Έχω και μακρύτερο κατάλογο, αλλά ε, θα τα πούμε και διμερώς αν θέλετε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Ευχαριστώ κύριο Πάσκο Κάτι να προσθέσω μόνο. Νομίζω ότι γνωρίζετε ότι όσο προχωρούν στην τεχνητή νοημοσύνη πιο προηγμένες χώρες, οι άλλες χώρες που δεν έχουν την ευκαιρία θα προσπαθήσουν να το αντισταθμίσουν με τα πυρηνικά όπλα. Παρόλο που είναι δαπανηρά και τα δύο, τελικά αυτό μπορεί να αποδειχθεί ότι θα είναι το όπλο του φτωχού το πυρηνικό. Και δεν μπορούμε να σκεφτούμε ε, να χαλαρώσει ή να μειωθεί το πυρηνικό κατόφλι. Ε, ίσως και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ευχαριστώ πολύ επικίνδυνα πράγματα, λέει η Πρόεδρος βεβαίως. Έχετε δίκιο. Τώρα έχει έρθει η ώρα των ευχαριστειών. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους εξαιρετικούς ε, ομιλητές μας. Μας βοήθησε πάρα πολύ ε, η παρουσία τους και η συνεισφορά τους στη τελευταία μας συνεδρίαση για την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο της Υποεπιτροπής ΣΕΝΤΕ Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ να χειροκροτήσουμε μαζί τους ομιλητές μας. Then allow me Και τώρα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλους εσάς για τις εξαιρετικές συζητήσεις που είχαμε και τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις. Οφείλω να πω ότι πραγματικά ε, το χάρηκα την ευκαιρία αυτή που είχα να προεδρεύω. Ε, κάτι που δεν περίμενα ούτε και εγώ, γιατί στην αρχή ήμουν πολύ διστακτική να αναλάβω, αλλά πραγματικά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που με βοηθήσατε να καταλάβω τη σημασία αυτή. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τη γραμματεία μας. Θυμίζω ότι είχαμε τρεις αλλαγές στη γραμματεία, τρεις επικεφαλής της γραμματείας. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για τη βοήθεια. Πάρα πολύ καλή η συνεργασία μας, όντως εξαιρετική και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είχαμε την ευκαιρία συνεχώς να ε, βασιζόμαστε ε, στην εξαιρετική γραμματεία μας. Και τέλος, χωρίς αυτό να είναι καθόλου το λιγότερο σημαντικό, θέλω να ευχαριστήσω τους διερμηνείς ήταν πραγματικά πολύ τεχνικές οι συζητήσεις μας ε, με λεπτομέρειες και πάρα πολύ ακριβή η διερμηνία. Σας ευχαριστώ πολύ.